Η σημερινή συνεδρίαση προβλέπει τα εξής στην ημερήσια διάταξη. Έγκριση της νομοδότησης του κυρίου Τσίτσεστερ, μια πρώτη συζήτηση ε, για την έκθεση της κυρίας Σόκεν, την ανταλλαγή απόψεων για τη διερευνητική επίστευση στην Ιταλία, για το θέμα που έχει να κάνει με τα απόβλητα, στις αναφορές έχουμε Τι αναφορές για τις γενικά τροπημένες οργανισμούς, για τα συμβάσει ορισμένου χρόνου εργασίας στα Ιταλικά σχολεία. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θα ήθελα να σας ζητήσω να εγκρίνετε τη σημερινή ημερησία διάταξη. Παρακαλώ, συνάδελφος Βαλέσσα. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την προσοχή σας ε, στο σημείο 18, στην αναφορά 18. Υπό το Β θα ήθελε η αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή το έχω αναφέρει αυτό στην γραμματεία και πιστεύω ότι δεν έχουμε εξαντλήσει τη συζήτηση για το θέμα αυτό και ότι θα έπρεπε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επί αυτής της αίτησης για το σημείο Β18. L'onorevole Sinclair. Sinclair. Thank you, Madam Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. παρατέταρτο έπρεπε να αρχίσει η συνεδρίαση αυτή. Έχουμε μισή ώρα καθυστέρηση. Έπρεπε να αρχίσει η ψηφοφορία σύμφωνα με την ημερήσια διάταξή μου 4 παρατέταρτο. Εγώ πρέπει 4 και τέταρτο να βρω κάποιον που ταξίδεψε 600 μίλια για να έρθει να με δει. Και δεν μπορώ να συμμετάσχω στην ε, ψηφοφορία. Γιατί δεν έγινε καθυστέρηση και γιατί δεν δόθηκε εξήγηση για την καθυστέρηση. Έχετε δίκιο, κυρία Σιγκλέρ. Ξέχασα να ζητήσω συγγνώμη από τους ε, παρόντες για την καθυστέρηση που σωρεύτηκε στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών που προηγήθηκε τη συνεδρία της Επιτροπής. Είχαμε μια διαδρομένη συζήτηση για ορισμένα θέματα που ήταν αντικείμενο της συνεδρίας των συντονιστών και έτσι λοιπόν δυστυχώς υπήρξε καθυστέρηση που δεν είχε προβλεφθεί. Ζητώ συγγνώμη και ζητώ από την κυρία Σινκλέρ ε, να ε, μην μας ζητήσει να αλλάξουμε την μερίσια διάταξη για την ψηφορία. Παρακαλώ. Να μπει στα πρακτικά αυτό. I have to leave to... Εγώ ήθελα να ψηφίσω και δεν μπορώ, διότι πρέπει να φύγω τώρα, πρέπει να πάω να βρω ένα πρόσωπο το οποίο ταξίδεψε 600 μίλια για να έρθει να με δει. Κυρία Σινκλέρ, ε, βεβαίω και γράφεται αυτό στα πρακτικά και ζητώ συγγνώμη. Επομένω. Ακούσαμε τι μα είπε και ο κύριος Βαλέσα για την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν αντιρρήσει ή μπορώ να θεωρήσω ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη για σήμερα. Γκρίνεται. Σημείο 2. Έχει μοιραστεί το έγγραφο που αφορά τις ανακοινώσεις για σχόλια. Υπήρξε κάποια απόκληση, αλλά έχει αποσυρθεί αυτό το σημείο. Δεν ε, βλέπω λοιπόν κάτι σε σχέση ε, με τις αμφιβολίες ε, που είχαν εκφραστεί στο παρελθόν. David Law mi ricordava che eh, abbiamo... Ο Ντέβιτ ε, μου υπενθύμισε ότι φιλοξενούμε μία αντιπροσωπεία Η, ε, από το Κανάρια, από την Ισπανία, που τον αδελφός Μάτο. Σας καλωσορίζω. Λοιπόν, τώρα, να σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των συντονιστών. Συνεδρίαση των συντονιστών για το πρώτο σημείο που έχουμε στην ημερησία διάταξη για τις διερευνητικές αποστολές για το 2013 αποφάσισε να εγκρίνει εν μέρη το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται επιλέχθηκε μία τροποποίηση για την εβδομάδα που προβλέπεται για την αποστολή στην Ελλάδα. Είχαμε ουσιαστικά θέση ως πιθανή ημερομηνία την εβδομάδα στην οποία πέφτει και πρωτομαγιά, όμως δεν θεωρήθηκε κατάλληλη αυτή η ημερομηνία, θα αναζητήσει άλλη εβδομάδα γραμματεία. Έτσι λοιπόν, κατόπιν ε, συζητήθηκε από τους συντονιστές η αναγκαιότητα να επαναοργανωθεί η αποστολή στην Πολωνία που ακυρώθηκε πριν λίγους μήνες επειδή δεν ήταν διαθέσιμα τα μέλη της αντιπροσωπείας. Επομένως, ε, περιμένει το Προεδρείο από τους συντονιστές μία πρόταση για το ποια μέλη θα συμμετάσχουν. Επίσης, κατόπιν ε, αιτήματος της κυρίας Βέρτμαν, ε, σε σχέση με τα αποτελέσματα της ε, εργασίας, της ομάδας εργασίας για το Λέιντε Κώστας, να ζητηθεί μία οργάνωση αποστολή στην Ισπανία για να μπορέσουμε να συναντηθούμε με τις Ισπανικές Αρχές για την ομοθεσία αυτή. Για τις, την ομοθεσία για τις παράκτιες ζώνε. Έτσι λοιπόν ζητήθηκε διαδικασία του κατοπήγοντο και θα ζητήσουμε από το Προεδρείο αυτή την άδεια. Επίση, κοινοποιώ σε όλα τα μέλη ότι στι 5 Δεκεμβρίου θα λάβει η χώρα το τρίτο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα άτομα με αναπηρία. Το φόρουμ αυτό θα, στο φόρουμ αυτό θα συμμετάσχουν και μέλη της Επιτροπής Αναφορών. Προβλέπετε δική μου παρέμβαση ως Προέδρου. Ε, προσκαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να συμμετάσχουν για το ζήτημα της οργάνωσης της ακρόασης για την ηθαγένεια που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου. Κοινοποίησα στους συντονιστές και θα σας πείσω και σε εσά ότι υπήρξε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έτοιμα να συμμετάσχει στην οργάνωση της ακρόασης και είναι αποδεκτό το αίτημα αυτό από τους συντονιστέ. Έτσι λοιπόν, πέρα από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, θα συμμετάσχει στην οργάνωση της ακρόσης και η Επιτροπή Γιούρη. Επίσης, υπήρξε συμφωνία επί της αναγκαιότητας να παρουσιαστεί στην Ολομέλη ένα ψήφισμα για το θέμα του Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Χάλιβα βάση της αναφορά Σίλβα, όμως δεν υπήρξε συμφωνία για την πρόταση του ψηφίσματος. Οι συντονιστές λοιπόν πρέπει να καταλήξουν σε ένα συμβασμό που θα έλθει εδώ στην Προεδρία και κατόπιν ε, εμείς θα δούμε όλο μέλο στο Στρασβούργο θα βάλουμε το ζήτημα. Η πρόταση του ΕΛΚ για την οργάνωση διερευνητικών αποστολών δεν συζητήθηκε. Η συζήτηση αναβλήθηκε για επόμενη συνάντηση για το έγγραφο που θα αφορά τους κανονισμούς που θα διέπουν την οργάνωση των αποστολών, η ομάδα των συντονιστών αποφάσισε να συνεισφέρει γραπτός προκειμένου να δοθεί μία ενίσχυση της θέσης της Επιτροπής Αναφορών στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ελήφθησαν άλλε αποφάσει από του συντονιστέ. και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θεωρούμε ότι εγκρίνονται οι αποφάσει αυτέ που ελήφθησαν. Να περάσω τώρα στο επόμενο σημείο της ημερικής διάταξης. Έχουμε αυτή την ε, αμφισβητούμενη ψηφοφορία για την γνωμοδότηση Τσίτσεστερ. Θέλετε το λόγο κύριε Τσίτσεστερ. Uh, uh, κύριε Πρόεδρε, καμία αντίρρηση να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Άρχεται ψηφοφορία. Να ψηφίσουμε. Τροπολογία, παράγραφος 1, ε, Μποστινάρου, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμό στην παράγραφο 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, παράγραφος 2, Μποστινάρου, καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε ο συμβιβασμός. Δεν ψηφίζουμε λοιπόν γι' αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την τροπολογία 3 και η τροπολογία 4 και 5 καταπίπτων γιατί έχει εγκριθεί ο συμβιβασμός. Τροπολογία 6 παράγραφος 3 Μπελιέ υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7, παράγραφος 3, άρου υπέρ. Κατά. We can check the vote with the machine. Να ελέγξουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Sorry, David. Vote 7. τροπολογία 7, 3, Δουλεύει. Six, six, one. No, no. No, no, we have, we have to, to, to open the vote. You already did. No? No. Start again, start again. Okay. Okay, we open... Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Κύριε Μποστινάρου, εντάξει. Ok. Va bene. It's okay. Anyone? No, there's one. We can close. Πέρασε. Six in favor, seven against, one abstention. Quindi l'emendamento è Απορρίπτεται. 8 παράγραφος 4 προς την Άρου. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Παράγραφος 4. Μπελιέ. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4. Τροπολογία 10. Κάτι. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξω. Άρχεται η ψηφοφορία για τροπολογία 10. Πέρας. Δέκα υπέρ, τέσσερις κατά. Γκρίνεται. Τροπολογία 11 στην παράγραφο 4. Βαλέσσα. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Γκρίνεται. Συμβασμός παράγραφος 5 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12, 13, 14, 15, όλες αυτές καταπίπτουν. Να ψηφίσουμε το συμβασμό 3 στην παράγραφο 6 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι τροπολογίες 16, 17, 18. Ψηφίζουμε την 19 για την παράγραφο 6α. Συνάδελφος Κολάρσκα Μπουμπίνσκα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 στην παράγραφο 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7, τροπολογία 21, μπελιέ υπέρ. Συγγνώμη, καταπίπτει, καταπίπτουν 21 και 22. καταπίπτει. Πρέπει να ψηφίσουμε την 22. 22. Περ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. Τροπολογία 23 στην παραγραφή 8. Μπελιά υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. Τροπολογία καταπίπτει 23, 25, παράγραφος 9, μπελιέ, υπέρ. Κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για την νομοδότηση, υπέρ. Κατά, εποχές, εγκρίνεται. Κύριε Τσίτσιστερ. Uh, uh, Κύριε Πρόεδρε, ε, εγώ εργάζομαι σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήθελα να σα πω ότι εάν κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία θα πρέπει και να γίνει και η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Προτείνω. Ναι, είναι ηλεκτρονικά θα γίνει πρώτα. Τελευταία ψήφο. Τελική ψήφο. Chiusa 13 υπέρ, 2 εποχές. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια κύριε Τζίτσαστερ. Ευχαριστούμε. Και πάλι κύριο Τζίτσαστερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. <laughs> Όποιος θέλει 13 είναι άτυχος. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τώρα τη διαδικασία της ψηφοφορίας, Να περάσουμε στην έκθεση για την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Μεσολαβητή για την έρευνα σχετικά με την προσφυγή κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Ουκέν είναι η συγγήτρια και έχετε το λόγο. Έγινε διεξοδική συζήτηση, λέει η κυρία Ουκέν. Να μην τα ξαναλέμε. Το κείμενο είναι μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Ήταν πάρα πολύ καλή η συνεργασία μας. και ξεκαθαρίζω ότι δεν ήταν θέμα του νέου 10 τη Βιέννη, απλώ δεν πρόκειται περί συγκρούσεω μεταξύ Διαμεσολαβητού και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, νομίζω ότι εξομολύθηκαν διαφορέ και τώρα πλέον δεν υπάρχουν ε, αντιπάθειε μεταξύ μα. Οι τροπολογίε θα ψηφιστούν 20 Ιανουαρίου του χρόνου. Grazie onorevole Oken Bostinaru. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, σας επιβεβαιώνω ότι σε αυτή την περίπτωση η εξαίρετη Μαργαρίτα ε, Άουκενε ενήργησε ως ειρηνοποιός, οπότε και τελικά επίσης αποσπάσαμε πάρα πολύ ε, σημαντική υποστήριξη για το σχέδιο κειμένου το οποίο προετοίμασε. Δεν μπορώ παρά να τη συγχαρώ την Μαργαρίτα, μια από η Επιτροπή μας και όλοι όσοι είναι πλάκοι μας σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης ε, καταφέραμε να δείξουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτός δεν είναι τρόπος να μπορεί να, να, να ενεργεί έτσι κάποιο θεσμικό όργανο. Είτε πρόκειται όταν συνομιλεί για το, με τον Διαβεσολαβητή, είτε όταν πρόκειται με κάποιο κράτος μέλος. Αυτό, αυτό, αυτό τονίζει τον θεσμικό μας ρόλο σε σχέση με τις ε, αναφορές του λαού. Γεια. βάλε τα ακουστικά. Παρακαλώ. Ο κύριος η ε, εισηγητής κύριος Μπέκερ, δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά μου είπε να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά. Είδες, μπορεί να γίνει συνεργασία καμιά φορά καλή και με τη δική μας την ομάδα και ο συνάδελφος Μπέκερ όπως ε, είπα ευχαριστεί θερμά για την καλή συνεργασία και θεωρεί επίσης ότι διαπιστώθηκε ότι τώρα δεν υπάρχει παραβίαση του ε, κειμένου ευρωπαϊκού δικαίου. Κάνει και κάποιες προτάσεις, αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο... Είναι βελτιωτικές προτάσεις και εν ώψη του χρόνου θα τις δώσω να συμπεριληφθούν γραπτώς στα πρακτικά. Υπάρχουν στην ομάδα... Ε, έχουν, έχουν ε, γίνει κάποιες ε, συνεννοήσεις και με την κυρία Όκεν ε, και με μας. Οπότε είναι καλή στιγμή αυτή για την Επιτροπή Αναφορών. Λαμβάνεται υπόψη η θέση του. Είναι καλή ώρα και για σένα και για την Επιτροπή όμως και για τους δύο. Σημαδιακή ώρα. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την, καταγγελία, την θέση του διαμεσολαβητή και είναι πολύ σημαντικό ότι ο τελευταίος προτείνει και διαδικαστικές βελτιώσεις, γιατί δεν πρέπει να διαπιστώνουμε μόνο ότι κάτι δεν πήγε καλά ή ότι κάτι πήγε όχι τόσο καλά, όχι. Θα πρέπει να κάνουμε και βελτιωτικές προτάσεις για να μην ξαναδημιουργηθεί πρόβλημα στο μέλλον. Έτσι πρέπει να εκλαμβάνουμε διαπαραταξιακά τη δουλειά στην Επιτροπή μας των Αναφορών, οπότε πολύ καλά πήγαν όλα. Ευχαριστούμε και την εισηγήτρια και τους σκιώδεις. Αυτά τα είπα ε, για λογαριασμό του συναδέλφου Μπέκερ. Ευχαριστούμε κυρία Βέρτμα, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι και εγώ θα συμφωνήσω και θα προσθέσω τις δικές μου ευχαριστίες εκείνες του συναδέλφους. Η κυρία Άουκεν απέδειξε ότι ε, έκανε εξαιρετική δουλειά και υπήρξε και υποδειγματική συνεργασία. Ευχαριστώ και από τη δική μου την πλευρά λοιπόν. Συμπέρασμα δηλαδή, αφήστε τα σε μένα. Τι ωραία να βλέπουμε τόση αρμονία στην Επιτροπή. Δεν υπάρχουν λοιπόν άλλε παρεμβάσει. Να υπενθυμίσω, όπω και η κυρία Όκεν, ότι η για την κατάθεση τροπολογιών είναι στις 12 Δεκεμβρίου. Το έγγραφο θα εγκριθεί στις 21-22 Ιανουαρίου και κατόπιν το Μάρτιο στην Ολομέλεια. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην πρώτη εντελεγή απόψεων για τη διερευνητική επέστρεψη στην Ιταλία. Θα δώσω το λόγο στην Αδερφή Μέρκης. Δεν είναι πρώτη φορά που πήγαμε στην Ιταλία για να δούμε αυτές τις πολιτικές και τις αναφορές για κατεπήγοντα για τα απόβλητα. Πήγαμε λοιπόν κυρίως λόγω των ανησυχιών των αναφερόντων, όχι μόνο από την περιοχή της Καμπανίας, όπου είχαμε κάνει προηγούμενη επίσκεψη πριν από δύο χρόνια, αλλά και από την περιοχή του Λάτσιο. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν και άλλες αναφορές που παρελήφθησαν από άλλες περιοχές, αλλά δεν πήγαμε σε αυτές τις περιοχές, παρόλο που ίσως επηρεάζονται από την ανικανότητα των πολιτικών αρχών να ε, πληρώσουν τις νομικές υποχρεώσεις τους για τη διαχείριση των αποβλήτων. Η προηγούμενη επίσκεψη ήταν τον Απρίλιο του 2010 και ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της έκθεσης μπορεί να επαναληφθεί και τούτη τη φορά. Ε, και όντως συμπεριλαμβάνεται στην έκθεσή μας αυτή τη φορά. Μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της επίσκεψης μας ενημέρωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την Ιταλία επιδιώκοντας κυρώσεις λόγω της αποτυχίας μετά τις διαδικασίες επί της Ιταλική, των Ιταλικών αρχών να εφαρμόσουν την απόφαση του δικαστηρίου από τον Απρίλιο του 2007. Και αυτό αφορούσε έλλειψη συμμόρφωσης με την κοινοτική νομοθεσία ε, για τις χωματερές, όπως ε, είπε η Κομισιόν πάνω από 255 χωματερές, ε, ε, από αυτές πολλές έχουν και επικίνδυνα απόβλητα. Ήταν πολύ επίκαιρη λοιπόν αυτή η επίσκεψη και συζητήσαμε το θέμα, μπορέσαμε δηλαδή να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Υπουργό Περιβάλλοντος της Ιταλίας. Είναι σαφές ε, ότι υπάρχουν πέντε πολύ σημαντικά θέματα και αυτά είναι, σημειώσαμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι αποτελεσματική παρακολούθηση δεν υπάρχει για να προληφθεί υπεραιτέρω, ε, το, το, το, περαιτέρω άνοιγμα παράνομων χρωματερών. Υπάρχει ενδημική αποτυχία η οποία πιάνει δεκαετίες ανικανότητας αντιμετώπισης των ε, αποβλήτων στην Ιταλία. Και αυτή η ενδημική αποτυχία έχει επιζήμια επίδραση στην υγεία του πληθυσμού που ζει κοντά στις μεγάλες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. Υπάρχει μεγάλη δομική ανεπάρκεια στο πολιτικό σύστημα της Ιταλίας που δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα και να λάβει αποφάσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής αποβλήτων. Υπάρχει και έλλειψη διαφάνειας και καθαρότητας ε, σε ό,τι αφορά την ευθύνη της λήψης, για τη λήψη των αποφάσεων. Ποιος είναι υπεύθυνος σε ποιο επίπεδο. Αυτή η ενδημική ε, αποτυχία οδήγησε στην υιοθέτηση κατεπίγουσας νομοθεσίας και στο διορισμό ειδικών νομαρχών, ειδικών επιτρόπων με εντολή να βρουν λύσεις στα κατεπήγοντα και στις κρίσεις των αποβλήτων ιδιαίτερα ε, στην Νάπολη και τη Ρώμη. Τώρα φαίνεται σαφέστατο ότι οι διορισμοί αυτοί και οι εντολές αυτές δεν συνάδουν με την ε, νομοθεσία της Ένωσης. Και πέμπτον, αυτές οι αποφάσεις επιβάλλονται στους ΟΤΑ και στις περιφερειακές αρχές χωρίς τοπικές και περιφερειακές αρχέ, σωτά, δηλαδή χωρίς διαβουλεύσει. Η τωρινή εθνική κυβέρνηση φαίνεται να καταλαβαίνει πολύ καλά την κατάσταση και είναι αποφασισμένη να αναδιοργανώσει τι πολιτικές δομές για να ανταποκριθεί στα θεμελιώδη θέματα που προανέφερα. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι υπάρχουν διαρθρωτικές αδυναμίες και οι οποίες είναι το χρόνο σιγά σιγά επηρέασαν και το οργανωμένο έγκλημα το οποίο διήθησε, διείσδησε σε αυτά τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Αυτή υπάρχει ειδική επιτροπή στην Ιταλική Βουλή η οποία συστάθηκε ειδικά για να εξετάσει τη σχέση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και της διαχείρισης των αποβλήτων ή τα εγκλήματα με τα απόβλητα. Ε, η Επιτροπή αυτή μάλιστα αυτή τη βδομάδα αντιλαμβάνομαι θα επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι καλό. Ένα ε, πρόσθετο πρόβλημα είναι και που γίνεται ακόμα πιο σοβαρό επειδή δεν υπάρχουν ε, πολλά δημόσια κονδύλια πιστώσεις είναι η κατανομή των οικονομικών πιστώσεων και πόρων. Φαίνεται ότι δεν επετεύχθη ευαρκής χρηματοδότηση ώστε να συμμορφώνεται η διαχείριση αποβλήτων με την κοινοτική νομοθεσία. Επίσης η Ιταλία πρέπει να διασφαλίσει ότι η ιεράρχηση των αποβλήτων θα τηρηθεί και ότι τα απόβλητα θα προλαμβάνονται κυρίως και θα μειώνονται επίσης σημαντικά και η διαλογή και η ανακύκλωση και η ανάκτηση ακολουθούν. Συνήθως όμως δεν φτάνουν ούτε στο στάδιο της σωστής διαλογής των αποβλήτων. Για πολλά χρόνια οι Ιταλικές αρχές δεν επένδυσαν αρκετά ούτε οικονομικά, ούτε αφιέρωσαν και μεγάλη προσοχή. Και έβρισκαν μόνο βραχυπρόθεσμες λύσεις με το φτηνότερο κόστος που οδήγησε σε αυξημένο μακροπρόθεσμο κόστος για την ε, Ένωση και την υγεία. Εμείς θέλουμε να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ε, συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία και σωστή ιεράρχηση και διαχείριση των αποβλήτων. Είδαμε ότι σε πολλές πόλεις, όπως την Νάπολη για παράδειγμα, Υπάρχει μια νέα ευαισθητοποίηση, μια νέα αρχή διαχείρισης των αποβλήτων. Είδαμε τα, να παρουσιάζονται προγράμματα διαχείρισης ε, αποβλήτων που είναι σωστά και συνάδουν και με την ενωσιακή νομοθεσία. Αυτό που κατέστη πρόδειλο και με οδυνηρό τρόπο είναι η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των κοινοτήτων και των αρχών. Υπάρχει πλήρης απουσία γόνιμου διαλόγου. Το έχουμε ξαναδεί αυτό σε προηγούμενες, ε, ε, σε προηγούμενες επισκέψεις από τον Απρίλιο του 2010 συγκεκριμένα και είδαμε ότι υπάρχει λίγος αμοιβαίος σεβασμός από τις αρχές προς τις κοινότητες και πολλές φορές και αντίστροφα από τις κοινότητες τους πολιτικούς. Και αυτό οδηγεί σε αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Νομίζω ότι πραγματικά ήρθε η ώρα και συμφωνήσαμε όλοι σε αυτό. Ήρθε η ώρα οι κοινότητες και οι αναφέροντες να εισακουστούν, να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί και να ακουστεί η φωνή τους, γιατί έχουν πολλά να συνεισφέρουν είναι πολύ σημαντική η συμβολή τους, αρκεί οι αρμόδιες αρχές να το καταλάβουν αυτό. Το ακριβές πρόγραμμα υπάρχει στην έκθεση ε, σε κάθε λεπτομέρεια, οπότε δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτών που είδαμε και δεν θα αναφέρω τους συνομιλητές μας. Γυρίσαμε φορτωμένοι με κιλά υλικού, αυτό είναι 7 κιλά που σας δείχνω εκεί. Και έχουμε κι άλλα. Ε, πλαστικό και έχουμε φωτογραφίες. Πολύ υλικό. Μη επεξεργασμένα απόβλητα εδώ, παράνομες χωματερές, όλα τα φωτογραφίσαμε. Έχουμε και DVD και φωτογραφίες, οπότε έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες και τεκμηρίωση που μας τις έδωσαν οι αρχές και οι αναφέροντες. Και με πολλή βοήθεια θα τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι είμαστε δύο επίσημα μέλη στην αντιπροσωπεία, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Μας συνόδευαν ε, οι Ιταλοί Ευρωβουλευτές, συνάδελφοι, που συνέβαλαν πολύ σημαντικά την ε, αντιπροσωπία μας. Επίσης αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη στην πολιτική και στις αρχές. Και ήταν ουσιώδης ο ρόλος τους γιατί πήγαν να συνδέσουν πάλι τις κοινότητες με τις αρχές. Τέλος πολύ σημαντικό, ο κόσμος ήταν παρόν. Όπου πηγαίναμε, συναντήσαμε πλήθη μεγάλα ανθρώπων πολύ αφοσιωμένων και ενθουσιωδών για τα θέματα αυτά. Μας ακολούθησαν στις ε, επισκέψεις μας και βέβαια δεν πρέπει να υποτιμήσουμε και τη συμβολή των αναφερόντων. Όλοι περιμένουν από την Ευρώπη να κάνει κάτι. Και αυτό είναι μεγάλη ευθύνη για μας. Κυρίως είναι μεγάλη ευθύνη για τις αρχές σε κάθε επίπεδο στην Ιταλία. Η κατάσταση στην περιοχή του Λάτσιο είναι κρίσιμη, εξακολουθεί να είναι κρίσιμη και φαίνεται, φάνηκε σε εμά τα μέλη της αντιπροσωπείας ότι η εθνική κυβέρνηση όχι μόνο γνωρίζει την κατάσταση, αλλά είναι διατεθειμένη να κάνει και κάτι. Και ο τωρινός Υπουργός Περιβάλλον είναι πολύ θετικός και επικοδομητικός και χρήζει και αξίζει την υποστήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την τεράστια αρνητική κληρονομιά. Είναι σαφές επίσης ότι ο ρόλος ε, του ειδικού επιτρόπου στο Λάτσιο δεν προσαρμόζεται καλά στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος εκεί υπήρξε κακοδιαχείριση επί δεκαετίες και αυτές οι ε, καινούριε ε, ε, πήγουσες αρμοδιότητες που δόθηκαν είναι αντιεπικοδομητικές και παραβιάζουν και την κοινοτική νομοθεσία. Και είδαμε και ένα θέαμα όπου διαφωνούσαν οι περιφερειακές και οι επαρχιακές αρχές και η μία έριχνε την ευθύνη στην άλλη σχετικά με το ποιος πρέπει να ε, εφαρμόσει την νομοθεσία για τα απόβλητα. Δεν επικεντρώνονταν σε αυτά που έπρεπε να κάνει ο καθένας, αλλά έριχνε ο Έλληνας την ευθύνη του στον άλλον. Αυτό δεν λύνει την κρίση. Το επίπεδο των δημοσίων διαβουλεύσεων είναι πολύ χαμηλό και στην περιοχή του Λάτσιο και ο ντόπιο πληθυσμό νιώθει ότι οι πολιτικέ αρχέ τον αγνοούν πλήρω. Η πολιτική για τα απόβλητα μέχρι τώρα ήταν πολιτική χωματερών και ακόμα και προσωρινών μετα... Ε, χωματερών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι πάνω σε αυτό το θέμα. Η αντιπροσωπεία είναι εναντίον οποιονδήποτε νέων χωματερών που θα υπάρχουν στο Ριάνο, πιάνουν τα Όλπο, Μόντε, Ντελακάρτσο ή όποιο άλλο σημείο. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προσωρινές. Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να παρέμβουν υπέρ τη ασφάλειας και του Μαλγκρότο για να μην γίνει άλλη βλάβη στην περιοχή, άλλη ζημιά. Τέλος, για να τελειώσω με την Νάπολη, συμφωνούμε με το Δήμαρχο της Νάπολης ότι η ιδιωτικοποίηση συνέβαλε στην καθοδική πορεία στην διαχείριση με καταστροφικές συνέπειες για τον τόπιο πληθυσμό και ωφέλησε μόνο την εγκληματικότητα που αυξήθηκε. Παράλληλα, δημόσιοι οργανισμοί θα πρέπει να είναι υπεράνω υποψίας, να δρούν με διαφάνεια και καλή διαχείριση. Αυτές είναι πολλές προϋποθέσεις και όροι που πρέπει να πληρούνται και αντιλαμβανόμεθα ότι η Αταλία αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση και σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο διαχείρισης. Εμείς στην Επιτροπή αυτή αναλαμβάνουμε πλήρη δέσμευση υπέρ των αναφερόντων αλλά και υπέρ των αρχών και των Ιταλών συναδέλφων για να βοηθήσουμε να υποστηρίξουμε ε, μια βραχυπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Όκεν. Δεν ε, θα μιλήσω για πολύ καιρό, για πολύ ώρα, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μέρκης ε, για την πολύ καλή συνεργασία. Ήταν πολύ δύσκολη αυτή η αποστολή. Είχαμε πάρα πολλή δουλειά, αλλά ήταν πολύ χρήσιμο αυτό το ταξίδι. Είχαμε ικανοποιητικά αποτελέσματα και θέλω να ευχαριστήσω και τους Ιταλούς συναδέλφους και κυρίως ε, κύριο την κυρία Τζελίλη που ε, μας βοήθησε στο να ενδυναμώσουμε την Επιτροπή και το αίσθημα ότι κάνουμε ομαδική δουλειά εδώ. Απλώς θέλω κάτι να προσθέσω στο είπε Όταν ήμασταν στην Άπολη, και συναντηθήκαμε και με το Δήμαρχο και με τον Υπουργό Περιβάλλοντος ε, της ε, Περιφέρειας. Ε, μπορώ να σας πω ότι σοκαρίστηκα γιατί μετά τη συνάντηση στη Ρώμη που μπορέσαμε να δούμε ότι ουσιαστικά το μπαλάκι το έστειλε ένα στον άλλο και κανένα δεν αναλάμβανε την ευθύνη. Λες και έπαιζαν μπάσκετ, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί παίκτες και ήταν αδύνατο να δούμε ποιος ήταν υπεύθυνο γιατί. Απλώς το μπαλάκι πήγαινε παντού. Αλλά κατόπιν όταν πήγαμε στην Άπολη και ακούσαμε ότι ο αρμόδιος υπουργό περιβάλλοντος ε, είχε 551 ε, δημαρχούς σε μία περιφέρεια. Τότε καταλαβαίνετε γιατί δεν λειτουργούν τα πράγματα. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε τόσο τεράστια συστήματα, μακροσυστήματα όπως βλέπουμε σε ορισμένες περιοχές, αλλά όλοι κατανοούν ότι ε, δεν ε, μπορούμε να έχουμε διαφάνεια σε μια τέτοια διοικητική δομή και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναφέρεται και στην έκθεση. Και η εντύπωσή μου ήταν αυτή όταν ε, μίλησα με τους Ιταλούς συναδέλφους, ότι γνωρίζουν ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και πρόκληση δηλαδή με το πώς είναι οργανωμένος ο δημόσιος τομέας. Και τώρα να σας πω ότι όσοι συμμετείχατε στις διερευνητικές επαστολές ε, πρέπει να συνειδητοποιήσετε πόσο σημαντική είναι η δουλειά μας όταν ε, συναντάμε τους πολίτες. Ακόμη και αν ε, είμαστε μια μικρή αποστολή, εκατοντάδες μας περίμεναν για μια μισή ώρα να φτάσουμε και μάλιστα παρέμειναν όταν έφτασαν και έτσι τους δίνουμε την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πιο σημαντικός δημόσιος φορέας, πιο σημαντικός δεσμός που τους παίρνει σοβαρά και τους σέβεται και ε, δεν τους αγνοεί. Και νομίζω ότι πρέπει να εκτιμήσουμε εδώ τη δουλειά που κάνουμε για τους πολίτες και οι διερευνητικές μας αποστολές ε, δημιουργούν ε, πολύ μεγάλο σεβασμό για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό ήθελα να το τονίσω. Ευχαριστώ κυρία Άουκεν. Να δώσουμε τώρα το λόγο στο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να μας παρουσιάσει και την άποψη της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Πολύ εκτιμούμε αυτές τις διερευνητικές ε, αποστολές, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου η Κομισιόν, όπως είπε και η κυρία Μέρκης, παραπέμπει στο δικαστήριο την Ιταλία για να επιβληθούν κυρώσεις. Το κάναμε αυτό πρόσφατα. Δεν αποκλείω να ξαναγίνει κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Και γι' αυτό θέλουμε να δούμε και εμείς αυτές τις πληροφορίες που φέρατε πίσω από την Ιταλία γιατί θα επηρεάσει τις αποφάσεις μας και τη συνέχεια που θα δώσουμε. Ευχαριστώ κυρία Αντζελίλη. Περίμενα να ακούσω κάποιο σχόλιο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή να αναφερθεί περισσότερο στην ουσία του κειμένου που λάβαμε σήμερα, τουλάχιστον εγώ σήμερα το διάβασα πρώτη φορά. Θα περιοριστώ λοιπόν σε κάποια σύντομα σχόλια. Αλλά πιθανότητα η πρόεδρος ίσως το έχει κάνει. Δηλαδή, ποια θα είναι η προθεσμία στο χρονοδιάγραμμα για την έκθεση αυτή. Σε ό,τι με αφορά, εγώ θα συνεισφέρω γιατί πιστεύω ότι ε, έχουμε ένα σημείο αφετηρίας, αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία που πρέπει να προσθεθούν στο κείμενο. Επίσης, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ιταλία λαμβάνονται αποφάσεις, γιατί στις 31 Δεκεμβρίου λίγη προθεσμία θα έπρεπε να κλείσει η Μαλαγκρότα στις 31 Δεκεμβρίου. ακούσαμε και κατά την επισκεψή μας, αναφέρθηκε και τώρα, για μια επιμήκυνση που θα μπορούσε να φτάσει μέχρι το Μάρτιο τον Απρίλιο, μια παράταση. Όμως, αντικειμενικά, η κατάσταση είναι πραγματικά επίγουσα. Και αναρωτιέμαι ποιο θετικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει αυτή η Επιτροπή προκειμένου να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια θετική λύση. Γιατί φυσικά οι πολίτες αναμένουν και ίσως και πολλά από την έκθεση αυτή. Και επομένως Ίσως μια επικοδομητική συνεισφορά θα έπρεπε να φτάσει από την δική μας Επιτροπή το συντομότερο. Αν και φυσικά γνωρίζουμε ότι το χρονοδιάγραμμα καθορίζεται από τη Γενική Ατζέντα. Πάντως οι πολίτες πραγματικά αναμένουν το συντομότερο μία έκθεση από την πλευρά μας. Ευχαριστώ κύριε Αντζελίλη. προτείνεται κάτι που δεν έκανα στην αρχή. Δηλαδή το σχέδιο κειμένο που συζητούμε σήμερα και οποίο θα έπρεπε να παρουσιαστεί στην οριστική του μορφή και θα έχει αμπλωτιστεί με τις συστάσεις που δεν υπάρχουν σήμερα στο κείμενο γιατί θα πρέπει να προκύψουν από μια συντονισμένη δουλειά και από τις ιδέες που θα προκύψουν και από τη σημερινή συζήτηση. Επομένως αυτό το οριστικό κείμενο θα πρέπει να παρουσιαστεί στην επόμενη συνεδρία του Ιανουαρίου. Η πρόθεση της Προεδρίας είναι να θέσει προθεσμία κατόπιν για τις τροπολογίες και να προτείνουμε ψηφοφορία το Φεβρουάριο. Και φυσικά ελπίζω να μπορέσετε να καταλήξετε σε κάποιου συμβασμού και σε μια συνεννόηση. Πάνω κάτω αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Δεν βλέπω να ζητά άλλο το λόγο. Επομένω, θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Μέρκη. Αν θέλει να κάνει κάποια καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για τη συνεισφορά σας κατά τη διάρκεια της αποστολής και για την παρουσία σας κυρίως ε, στην Καμπανία. Και επίσης ευχαριστώ και την κυρία Λτζελίλη που ήσασταν ε, παρούσα, σας ευχαριστώ και σήμερα για τη δεσμευσή σας. Προκειμένου να επανέλθω σε σας κυρία Όκεν. Σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία εκ νέου. Τον Απρίλιο του 2010 παρακολουθούμε το ζήτημα Είδαμε ότι το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικό στο ζήτημα αυτό, κυρίως λόγω των προσδοκιών των πολιτών, που είναι πάρα πολύ ψηλέ, πράγματι. Αυτό είναι αμφισβήτητο. Νομίζω ότι η απλή παρουσία μας ήδη κατι δείχνει, αλλά το είδαμε αυτό και την περασμένη φορά πάρα πολύ διεθνής βοήθεια κατέφτασε. Επίσης είδαμε ο υπουργό ε, να προσπαθεί να αλλάξει τώρα την τελική νομοθεσία προκειμένου να υπάρχει διαπεριφερειακή υποστήριξη. Ενώ στο παρελθόν έπρεπε να σταλίνονται τα απόβλητα στο εξωτερικό, εκτός Ιταλίας, για να αποτεφρωθούν. Και τώρα προσπαθεί ο υπουργό να το αλλάξει αυτό για να λύνεται το πρόβλημα εντός Ιταλίας. Και φυσικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαρίστω ε, να ανταλλάξουμε την τεκμηρίωση και ας κάνουμε κάτι για το περιβάλλον και πράγματι αυτό είναι ένα προκαταρκτικό σχέδιο μόνο. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ε, πρέπει να διαβουλευτούμε περαιτέρω, όχι μόνο με τα παρόντα μέλη, αλλά και με ε, δεν είναι παρόντες και να προσθέσουμε και περαιτέρω πορίσματα στην έκθεση για να ψηφίσουμε το Φεβρουάριο. Ευχαριστώ και πάλι κυρία Μέρκης. Θέλω να ευχαριστήσω και τη γραμματεία, λέει κυρία Μέρκης, για όλη τη τη βοήθεια. Και κατά τη διάρκεια τη αποστολή, αλλά και στη συνέχεια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμεί τη γραμματεία. Κλείνουμε το σημείο αυτό και να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινή διάταξη, που είναι η αφορά 338-2010 που παρουσιάστηκε από κάποιους Ισπανούς πολίτες ε, εξ ονόματος της πλατφόρμας για την υπεράσπιση των πράσινων κοιλάδων και έχει να κάνει με τη συλλογή δάτων και τη διάνοιξη γεωτρήσεων στο φυσικό πάρκο Σιέρα Κασόρλα. Ε, είναι παρόν για την αναφορά αυτή ο κύριος Γκαλβεσβία, τον οποίο δίνω το λόγο για πέντε λεπτά. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντα σα που μου αυτή την ευκαιρία σήμερα, ούτω ώστε να μιλήσουμε για μια φορά εδώ στο Κοινοβούλιο. Σα υπενθυμίζω ότι από το 2010 έχουμε υποβάλει αυτή την αναφορά στο Κοινοβούλιο για κάποιο είδου για αυτές τις γεωτρήσεις που γίνονται στο φυσικό πάρκο του, της καθόλου Las Vegas. Πρόκειται για μια ζώνη που προστατεύουν από διάφορε ε, οδηγίε και, δεν πάση περιπτώσει, πρόκειται για μια περιοχή κοινοτικού ενδιαφέροντο. Τον Μάιο, την ίδια χρονιά, είχαμε την ευκαιρία εδώ στο Κοινοβούλιο τη Επιτροπή σα να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μα ενημέρωσε για το ότι θέλει να αρχίσει μια διαδικασία επί παραβάση, λαμβάνοντα υπόψη το τι είχε γίνει. Και γιατί ισχυριζόντουσαν ότι έχουμε εδώ παραβίαση τριών οδηγιών το Κοινοβούλιο επίση ετώνησε ότι θα πρέπει με πήγοντα χαρακτήρα να ενεργήσουμε και είπε ότι πρόκειται για κάτι το οποίο είχε να κάνει με το περιβάλλον. Και όπω ορίζει η σχετική οδηγία, πρόκειται εδώ πέρα για την τήρηση του δικαιώματο του, τη υποχρέωση σοφροσύνη και προσοχή. Γιατί είχαμε πάλι πολύ σημαντικέ ζημίε που είχαν προκληθεί. Συνεχίζονται οι ζημίε. Ε, ξεκίνησε η υπόθεση από τον Μάιο, εδώ και 7 μήνε περίπου. Ε, και το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτή την μαζική γεώτρηση. 45 λίτρα το δευτερόλεπτο ήταν η άδεια που είχε δώσει η κυβέρνηση. Και από Μάιο μέχρι Οκτώβριο, επί 7 ώρες, επί 12 14 ώρες Δηλαδή έχουν αντιληφθεί από αυτό το φυσικό πάρκο σε αυτήν την προστατευόμενη ευρωπαϊκή περιοχή, γιατί ε, μιλούμε εδώ πέρα ε, για το ισοδύναμο δύο Ολυμπιακών πισινών. Ολυμπιτήριο. Παρά λοιπόν τα, τις ενστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ τώρα έχουμε ε, αποξήρανση, έχει, έχει, έχει, έχει ε, αποψηλωθεί ούτως ε, υδροφός ορίζοντας και οπότε. Εδώ συνεχίζεται το πρόβλημα και το θέμα είναι εμεί ω πολίτε τι, τι μπορούμε να πούμε. Τι θα πούμε δηλαδή στον κόσμο, γιατί έχουμε 7 μήνε που περάσανε. Είναι απαράδεκτο ότι δεν έχει αρχίσει ακόμα αυτή η διαδικασία η παραβάση του τη Ευρωπαϊκή Οπότε γι' αυτό και ελπίζουμε ότι αυτό το μέτρο το οποίο είχε ε, ε, ανακοινωθεί θα, θα γίνει με τη εκπαιδευτική ε, ταχύτητα που μα έχει στο Κοινοβούλιο. Και σα υπενθυμίζω ότι συνεχίζονται αυτέ οι γεωτρήσει με τι συνέπειε που σα περιέγραψα. Τώρα, χωρίς να μακρηγορώ, θα πρέπει να σας αναφέρω το ότι εμείς προσδοκούμε το ότι αυτό το οποίο πρέπει να, να, να ξεκινήσει η Κομισιόν ή είναι ότι ένεξη της διαδικασίας ή παραβάσει ούτως ώστε οι Ισπανικές αρχές να λάβουν τα μέτρα τα οποία επιβάλλεται ε, επί τη βάση του γενικού δικαίου και η λύση η οποία θα δοθεί να είναι ε, τέτοια ούτως ώστε να υπάρξουν εγγύησεις ούτως ώστε η οικολογική αξία ε, της περιοχής να αναδειχθεί, να προστατευτεί όπως ορίζουν αυτές οι τρεις ε, οδηγίες τις οποίες λέει η Κομισιόν ότι τις έχει παραβιάσει αυτή η δραστηριότητα και επίσης η λύση επιδιωκόμενη να είναι τέτοια ούτως ώστε αυτού του είδους υγειοτρήσεις να μην γίνονται στο πάρκο αυτό, σε αυτή την περιοχή, να γίνεται απ' έξω, έξω. Και έτσι, οικολογικά να μην πλήσει την περιοχή. Οπότε, αυτό που έκανα και εγώ, να μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Δηλαδή, κανείς να πάει στην σελίδα Ευρώπη να δει τι ε, τις, τις σχετικές καταχωρήσεις για το Natura 2000 και ε, να μπορεί λοιπόν ο κάθε πολίτη να ενημερωθεί. Γι' αυτό και σας λέω ότι τα κείμενα αυτά και οι στάσεις για την εφαρμογή των οδηγιών εμένουν στο ότι θα πρέπει αυτές τι δραστηριότητε να μην γίνονται σε προστατευόμενη ζώνη. Επίσης, παρακαλώ να μην ξεχνάτε ότι αυτές οι εξωτερικέ δραστηριότητε μπορεί να έχουν επιπτώσει όσον αφορά την πανίδα και χλωρίδα της με μέσα στη συμπληρωτευόμενη ζώνη και ας γίνονται δραστηριότητες εκτός. Άρα χρειάζεται να υπάρξει απόκριση άμεση από τα κράτη-μέλη, από την Κομισιόν και, εν πάση περιπτώσει, να προστατευτούν τα κοινοτικά συμφέροντα. Και η λύση να είναι τέτοια ούτως ώστε να προστατεύεται η ακεραιότητα αυτή τη προστατευμένη περιοχή και να μην έχουμε εμβαλωμετικές λύσει, οι οποίε οδηγούν στο να συνεχίζεται η επιζημία δραστηριότητα όπω έγινε του τελευταίου μήνε. Και ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ και επειδή σεβαστήκατε και το χρόνο. Τώρα ο πρόσωπος Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι. Τον Μάιο. Ήρθαμε εδώ και σας είπαμε ότι θα αρχίσει, αρχίζει η διαδικασία η παραβάση επί τη βάση των πραγματικών περιστατικών που αναφέρει αυτή η αναφορά. Και αυτό διότι εδώ πέρα υπάρχει ισχυρισμό παραβιάσεως του κοινωτικού δικαίου. Δεν ευδοκίμησε η μελέτη των επιπτώσεων αυτών των γεωτρήσεων σε σχέση δηλαδή με τη, τη, λεκάνη των τροφόρων ορίζοντα ε, τη, τις λεκάνες απορροής κλπ. Και επίσης όπως είπε και ο αναφέρον ή αναφερόμενος, έχουμε τα διαδήματα που αρμόδιες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, και όσο αργότερα, τον Ιούνιο συναντήσαμε τις πανικές Αρχές και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μας πούν τι μέτρα έχουν υπόψη να λάβουν ούτως ώστε να πάψει η επιζημία δραστηριότητα. τώρα. Ίσως δεν είναι αγώγιμη αυτή η παραβίαση του κοινωτικού δικαίου. Απλώς, ίσως, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι, χωρίς άλλα μέτρα, χωρίς τη διαδικασία παραβίαση, να θέσουμε τέρμα εις αυτή τη δραστηριότητα. Ήρθαμε επομένω σε επαφή με τις Ισπανικές Αρχές και αυτή μας ε, διευκρινήσε αυτά τα οποία ζητήσαμε τον Ιούλιο. Επίσης, Αργότερα, το Σεπτέμβριο, ζητήσαμε ενημέρωση επιπλέον. Έγινε ενημέρωση από τον αναφέροντα και σε δέκα μέρες τις είχαμε. Οπότε με όλες αυτές τις πληροφορίες εμείς υποχρεούμε θα τις λάβουμε υπόψη να κάνουμε την αξιολόγηση αυτών των πραγματικών περιστατικών και τότε να αρχίσουμε τη δικασία παραβάση απευθύνοντα σχετική επιστολή στο κράτο μέλο. Και αυτό χρειάζεται, διότι εάν δεν το κάνουμε αυτό, αυτό θα είναι επιζήμιο για την συνέχιση της παραπέρα διαδικασίας. Πάντω θα πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να κάνουμε την ανάλυση και έχουμε λάβει τι τελευταίε πληροφορίε, μόλι από 10 μέρε. Οι ισπανικέ αρχέ είπαν ότι η Κοφεντεραθιόν Γεωγράφη είναι η αρμοδία Επιτροπή, η οποία ανέφερε στο Ισπανικό Συμβούλιο Γεωλογία και Εξορίξεων μια μελέτη, τόσο ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να είναι δυνατόν να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα, γιατί ακριβώ αν υπάρχει σχέση αιτίου αποτελέσματο μεταξύ τη γεωτρήσεω και των ενδεχομένων ζημιών που έχουν ε, επιφερθεί ει τον οικότοπο αυτό. Και στη συνέχεια δούμε τι λύσει είναι δυνατόν να έχουμε, τόσο ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια θεωρούσαν οι Ισπανικές Αρχές ότι όντως υπήρχε επιζημία δραστηριότητα αλλά δεν μπορούσαν ακόμα να δουν κατά πόσον υπάρχει μεταξύ γεώτρησης και ζημίας σχέση αιτίου αποτελέσματος. Και ακριβώς η μελέτη εις αυτό αφορούσε. Έγινε η μελέτη, ε, κοινοποιηθήκε σε εμά και είπαμε ότι από τη μια μεριά οπωσδήποτε υπάρχει κάποιο είδους ε, σχέση άμεση μεταξύ της γεώτρησης στην πηγή Μαγίγιο και των ζημιών που έχουν ε, ε, γίνει ε, τον οικότοπο. Όπως και σε άλλες και σε άλλες πηγές έχουμε κάποια προβλήματα. Εκεί όμως είναι πιο λιγότερο ξεκάθαρα τα θέματα. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Χρειάζεται επομένω μια σειρά από αναλύσεις και από μελέτες που πρόκειται να γίνουν. Επίσης, έχουμε ένα σωρό διορθωτικά μέτρα στην, διάμεσο διάστημα με, πριν γίνουν οι πλέον μελέτες και έτσι έχουμε πάυση της άντλησης ε, των υδάτων κατά την ε, ε, θερινή περίοδο. Έχουμε κάποια όρια, έχουμε κάποιες πηγές, κάποια κατόφυλλα τέλο πάντων που δεν μπορούμε, δεν μπορούμε αυτά να τα παραβούμε ούτως ώστε ε, να γίνεται η άντληση των υδάτων, η γεώτρηση και η συνομοσπονδία, η γεωγραφική για τον Κοδελκυβίρ είπε ότι πρέπει να λυθούν τα εξή μέτρα. Πρώτα πρώτα. Κατά την θερινή περίοδο, δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο, να έχουμε κάποια μέτρα, ώστε να σταματήσει αυτή η επιζημή δραστηριότητα. Και είπαμε αυτό προσωρινά μέχρι την ολοκλήρωση των, των συμπληρωματικών μελετών. Επίσης, ένα δεύτερο μέτρο που έχει προταθεί. Να έχουμε πρόγραμμα παρακολούθησης όσον αφορά τον τροφολογικό ορίζοντα για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Αυτό θα γίνει, γίνει συγγνώμη, από τον Ιούνιο του 2013, 12 ε, και μέχρι τον Μάρτιο του 2013 τρίτο μέτρο, το οποίο αφορά το να μελετηθεί ποιε μπορεί να είναι οι εναλλακτικέ όσον αφορά κάποιο σύστημα εκμετάλλευση, αλλά ακόμη ε, τα οριστικά συμπεράσματα συζητιά με αυτήν την εναλλακτική δεν μα έχουν ανακοινωθεί. Και έτσι να καταλήξουμε σε κάποια οριστικά μέτρα, να δούμε ακριβώ ποια είναι τα σημεία τη γεώτρηση και να έχουμε ε, τέλο πάντων ε, αλλαγή των υδρολογικών πόρων από αυτό που γίνεται με άλλους και να δούμε πώς θα αλλάξει η περιοχή η οποία ιδρεύεται και με κάποια ασφαλιστικά μέτρα να σταματήσει η δραστηριότητα της άντλησης των υδατών. Όλα αυτά εμείς θα μελετούμε με ρυθμού ταχύ σε σχέση με τον όγκο των πραγματικών περιστατικών που μας έχουν διαβαστεί. Ελετούμε τα υπέρ και τα κατά των μέτρων που προτείνει η Ισπανία και να δούμε πώς τελικά θα λυθεί το πρόβλημα, πώς θα σταματήσει να θεσμίζουν δραστηριότητε, τέλος πάντων θα υπάρξει νέα φουρνιά από τις δραστηριότητες. Τέλος πάντων. Αυτό το οποίο είχε προκύψει είναι ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο είναι νόμιμο όσον αφορά την διόντρηση για σκοπούς ποτίσματος πέρασε από αυτή την έγκριση χωρίς να έχει γίνει μια μελέτη για τις οικολογικές ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτής της δραστηριότητας. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χρειάζεται μια εκ των προτέρων αξιολόγηση Όταν όμως έχει διαπιστωθεί ότι αυτή η δραστηριότητα για τουλάχιστον ένα σημείο αναμφίβολα προκύπτει ότι υπάρχει ζημία και έχουμε όλες αυτές τις μελέτες τις πληματικές μελέτες τότε θα πρέπει να σταματήσει αυτή η δραστηριότητα. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί το να συνεχιστούν οι γεωτρήσεις είναι κάτι που δεν συνάδει προς την οδηγία Habitat σχετικά με την αρχή της πρόληψης και διαφύλαξης. Οπότε, σε περίπτωση αβεβαιότητας όσον αφορά τις πιθανές ζημίες που προκαλούνται. Άρα, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα της γεώτρηση. Και αυτό το, να, το να διαπιστώνεται πριν αρχίσει δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν μπορούν οι αρχές να είναι βέβαιες σε σχέση με αυτό, ούτω ώστε κανεί να αποκλείσει την επιζήμια ε, συνέπεια, τότε έχουμε ως συμπέρασμα ότι είναι, αν όχι βέβαια, είναι τότε πιθανή η ζημία στο περιβάλλον. Άρα εδώ συντρέχει το άρθρο 6.3 και 6.4 της οδηγίας. Σύμφωνα με τους τον από τον Μάιο, θεωρούμε ότι επί τη βάση των όσων μας είπαν οι αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να συνεχίσουμε την διαδικασία της προσφυγής επί και να διεκπαιρεώσουμε την υπόθεση όσο μπορούμε καλύτερα. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό ο κύριος Μιράντα. Η κυρία Μιράντα, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η παρακολούθηση της αναφοράς που, όπως είπε η Επιτροπή, ε, την απασχόληση καταρχήν τον Μάιο κατόπιν των επαφών με με τις ισπανικές αρχές της αυτόνομης περιφέρειας και των άλλων συναρμοδίων έδειξε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις κυρίως για το ότι έχουμε εδώ και πάλι παραβίαση της οδηγίας Habitat. Όλο προφάσεις είναι η Ισπανική κυβέρνηση και όλα αυτά που μετέρχεται, αλλά και εμείς θέλουμε να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ πέρα το timing έχει μεγάλη σημασία. Πιέζει ο χρόνο για την υπόθεση αυτή. Και τι διαπιστώνουμε. Ότι ενεργεί με βραδίτε το Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να ξεκινήσει τη διαδικασία η παραβάση. Επομένως, θα πρέπει δυναμικά να επιμείνουμε ούτως ώστε να έχουμε τους αναγκαίους μηχανισμούς ούτως ώστε να κινηθεί αυτή η διαδικασία. Επί τη βάση επομένω τη σχετική τεκμηρίωση, ε, και επί τη βάση των πληροφοριών που παρεσχέθησαν τον Αύγουστο του 2012, επί τη βάση του εγγράφου που έχω στα χέρια μου τουλάχιστον, δεν ξέρω μήπως έχουμε κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, διαπιστώνω από αυτά τα οποία εγγράφος υπέβαλε η Ισπανία του 2012 είναι ότι έχει νηθεί μια διαδικασία. Ούτω ώστε να έχουμε άντληση ενό λίτρου ανά δευτερόλεπτο στην πηγή μαγείλια. Αλλά από την άλλη μεριά τι έχουμε. Είχαμε αυτά τα 45 λίτρα ένα δευτερόλεπτο. Τα οποία στην πράξη αντλούν. Αυτό είναι σαν αστείο. Μάλλον αυτό δεν είναι ένδειξη θέλησης για να επιληθεί το πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν, έχουμε κάποιο είδους ε, πρόγραμμα, πλάνο, σχέδιο παραγωγή μέχρι τα μέσα 2013 και θα πρέπει όμως να ληφθούν και κάποια σοβαρά μέτρα προστασίας επί τη βάση αγροσαρκής προφύλαξης όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απλώς θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει εν αυτής κατάστασης είναι το ότι εδώ έχουμε σοβαρή βλάβη και του περιβάλλοντος εκεί στην οροσυρά καθόλου και θα πρέπει πιο προσεκτικά να μελετηθούν τα δεδομένα. Επομένως, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι δηλαδή αμελητή θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία παραβάση. Ε, να μην φτάσουμε στο σημείο που να είναι ανέκλητη βλάβη. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά άλλο το λόγο. Έτσι λοιπόν θα, έλεγα και, θα δίνω και πάλι το λόγο στον αναφέροντο για να απαντήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να απαντήσω στον ε, κύριο Βουλευτή ε, που μόλις έλεγε το λόγο ότι σύμφωνα μαζί του το να φερούμε το ότι έχουμε ε, μία ενίσχυση ουσιαστικά ε, νερού με ένα λίτρο ένα δευτερόλεπτο όταν η άντληση που επιτρέπεται είναι 45 λίτρα το δευτερόλεπτο είναι πραγματικά κακόγουστο αστείο. Δεν είναι ένα, πραγματικά ένας κατάλληλος τρόπος να απαντήσει η Ισπανική Αρχή σε ένα τόσο επίγον θέμα το να λαμβάνουμε μέτρα και το να συνεχίζουμε να κάνουμε αναλύσεις είναι κάτι που ελπίζαμε ότι θα είχε γίνει από πριν και το να συνεχίσουμε να το αναβάλουμε αυτό μέχρι το Μάρτιο μας ανησυχεί, γι' αυτό είμαστε εδώ και επιμείναμε και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε. Παρ' όλα αυτά χαίρομαι που άκουσα τις πληροφορίες της Κομισιόν σύμφωνα με τις οποίες ε, εξακολουθεί να θεωρεί τη διαδικασία επιπαραβάση ω κάτι απαραίτητο και άκουσα προσεκτικά τα λόγια της Επιτροπής όταν λέει ότι αυτή η διαδικασία περιβάσει θα επιδοθεί πολύ σύντομα. Ελπίζω να γίνει κάτι τέτοιο και ελπίζω ότι σε πολύ περιορισμένο χρόνο θα μπορέσουμε να βρούμε μια οριστική λύση για αυτή την περιοχή η οποία πραγματικά βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό κίνδυνο. Και τέλος, να αναφερθώ σε ότι υπόθηκε στην αρχή ότι η λύση πρέπει να είναι ικανοποιητική. Οι Ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν στις Ευρωπαϊκές αρχές και εμείς λάβαμε σχετικό αντίγραφο. Ανακοίνωσε το μεταξύ των πιθανών μέτρων είναι αυτοί να ε, σκεφτούν ε, να γίνουν αλλού οι γεωτρήσεις. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω ότι η λύση της μεταφοράς της τοποθεσίας σε άλλη περιοχή εκτός του πάρκου θα μπορούσε να είναι μια ευγενής λύση για να επιληθεί ένα πρόβλημα, όμως εγώ νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό που λέει ε, το ίδιο Ευρωπαϊκό Θεσμός, ε, τα ίδια τα ευρωπαϊκά όργανα, ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι μέτρα τα οποία μπορεί να εφαρμόζονται εκτό, αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι η συνέπεια εντό τη προστατευόμενη ζώνη. Ο στόχο πρέπει να είναι να καταργήσουμε οποιαδήποτε, να εξελίψουμε οποιαδήποτε περιβαλλοντική ζημία σε μια προστατευόμενη περιοχή που είναι πάρα πολύ σημαντική από περιβαλλοντική σκοπιά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για τη συνεισφορά που μας έδωσε. Είναι πάρα πολύ σε αυτή η έκθεση και υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση από ό,τι βλέπουμε. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει και γραφειοκρατία και ουσιαστικά βλέπουμε να υπάρχει μια απέτηση από τους ε, πολίτες, επομένως ε, από εμά ε, είναι σημαντικό να ακούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκει χρήσιμη τη συνεισφορά των πολιτών κυρίως, οι οποίοι διαμέσω ημών απευθύνουν απευθύνονται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι πάρα πολύ που στην περίπτωση αυτή ακούστηκαν ενδιαφέρουσες ιδέες. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από το να διατηρήσουμε την έκθεση νυχτή όπως αναφέρθηκε αλλά φυσικά θα προσπαθούμε να παρακολουθούμε και την κατάσταση και εμείς ε, φυσικά θα απευθυνόμαστε από την πλευρά μας στις Ισπανικές Αρχές αλλά και στην Κομισιόν θα τη ζητήσουμε πέρα από την αυστηρή στάση που θα πρέπει να έχει να ασκήσει και μεγαλύτερη πίεση για να επιταχύνει τους χρόνους επίλυσης της υπόθεσης αυτής. Ευχαριστούμε λοιπόν που μας παρουσιάσατε αυτή την αναφορά και να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο που είναι η αναφορά 813-2008. Έχει παρουσιαστεί από τον κύριο Τζον Μπράιαν η αναφορά αυτή. Σας δω συγγνώμη, αλλά τώρα λαμβάνουμε κάποιες θα συζητήσουμε ξεχωριστά, παρόσα όσο λέγονται στην μερική διάταξη, τις ε, αναφορές που έχουμε στο σημείο 10 και θα ξεκινήσουμε με την 813-2008 του κ. Brian Τζον και θα του δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ξαναμιλήσω. Ανησυχώ γιατί το πάνελ της ΕΦΣΑ για τους μεταλλαγμένους μικροοργανισμούς ε, παίρνει αποφάσεις που επηρεάζουν την υγεία εκατομμυρίων το, η κοινή γνώμη δυσπιστεί όμως ε, και απογοητεύομαι γιατί η Κομισιόν έδωσε συγκατάθεση για τα μεταλλαγμένα παρά τα προβλήματα στην υγεία θηλαστικών και ανθρώπου. Η ΕΦΣΑ και η Κομισιόν επίσης αγνόησαν την εχθρότητα της κοινή γνώμης προς τα τρόφιμα αυτά τα μεταλλαγμένα που ε, συγκέντρωσαν 1,2 εκατομμύρια υπογραφές ε, υπήρξαν λάθος επιστημονικές μεθόδους από την ΕΦΣΑ για τις ποικιλίε των μεταλλαγμένων και δεν ε, ε, χρησιμοποίησαν αναπαραγώγημα ε, πειράματα. Υπάρχει μια προκατάληψη υπέρ των μεταλλαγμένων στην ΕΦΣΑ. Δεν έκανε τίποτε η ΕΦΣΑ για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες μας αν και έγιναν κάποιες προσπάθειες στον τομέα πολιτικών και κανονισμών. Ο καθηγητής Σεραλίνη και άλλοι πρόσφατα δημοσίευσαν μια μελέτη για την τοξικότητα και τις ε, ζωοτροφές και ε, έδειξαν ότι είναι τοξικά αυτά, αυτές οι ουσίες στους επίμιες, στους όταν μπουν σε μικρές ποσότητες. Δεν, ε, υπήρξαν, δεν υπήρξε σύστημα συναγερμού ενώ υπάρχει ένα διετές ε, πείραμα που έγινε με, διάρκεια, ε, ε, με υψηλά πρότυπα ε, συνοψίζομαι ότι είναι ε, υψηλής τοξικότητας σε οργανισμούς μη στόχο, επηρεάζονται τα κύτταρα, μειώνεται η ε, αναπαραγωγική ικανότητα, ζωτικά όργανα καταστρέφονται. Αυτά είναι προβλέψιμα αποτελέσματα καλά καταγεγραμμένα, ενώ οι Κομισιόν και η ΕΦΣΑ συνεχώς κοφεύουν. Ε, όταν δημοσιεύτηκε το κείμενο Σεραλίνη, είπαμε να εξεταστεί πολύ προσεκτικά, να υπάρξει μορατόριουμ στις ε, εγκρίσεις και να επαναληφθεί, αν χρειαστεί, ένα πείραμα από την ερευνητική ομάδα και να ζητηθεί από την ΕΦΣΑ να ξαναδεί παλιές γνωμοδοτήσεις για, το, για τα μεταλλαγμένα, ιδιαίτερα για αυτές τις ουσίες που εξετάζουμε τώρα. Ε, λαμβάνοντα υπόψη τα ερευνητικά αποτελέσματα σε Ραλίνη. Ζητήθηκε γνωμοδότηση από την Κομισιόνα για το, την έρευνα Ραλίνη. Τώρα η ΕΦΣΑ εξέδωσε τι επόμενε εβδομάδε και άλλε γνωμοδοτήσει, λε και δεν είχε γίνει τίποτα. Και στι 18 Οκτωβρίου, ένα μήνα μόνο μετά τη δημοσίευση τη νέα έρευνα, η Κομισιόν έδωσε έγκριση για την αγορά για την, το μεταλλαγμένη αυτή ε, ε, εκδοχή του αραβόσιτου. Αυτό δείχνει ότι η Κομισιόν και η ΕΦΣΑ έχουν εγκαταλείψει τελείως την αρχή της προφύλαξης, παραβιάζοντας τις οδηγίες ε, και ακολούθησαν χειρότερα. Όπως είπαμε στην επιστολή μας στην Επιτροπή Αναφορών τον Οκτώβριο, η ΕΦΣΑ απάντησε άμεσα σχεδόν στην έρευνα σε Ραλίνη ε, από την αρχή ε, καταδίκασε την έρευνα και του συγγραφείς, έκανε και μια ενδιάμεση αξιολόγηση η οποία ήταν ε, τελείως ανάρμοστη, έκανε κάποιες επιστημονικές παρατηρήσεις αμφίβολες που απαντήθηκαν αμέσως από τους ερευνητές. Επίσης κάνει υποκριτική κριτική, λέει ότι δεν ακολουθήθηκαν πρωτόκολλα εργαστηρίων που αυτό δεν το ε, ζήτησε από τις μελέτες της Μονσάντο βέβαια. Επίσης ε, ζήτησε πλήρες σειρές, σειρές δεδομένων από τη γαλλική ομάδα ενώ ε, από τη Μονσάντο δεν τα ζήτησε. Ακόμα χειρότερο. Φάνηκε ότι η ΕΦΣΑ είχε φτιάξει μία task force πολύ, το, πολύ επιστημονική για να καταδικάσει την έρευνα Σεραλίνη και υπήρχαν και ε, δημόσιοι λειτουργοί με σύγκρουση συμφερόντων πολλές φορές έκαναν μια τηλεδιάσκεψη δε με επιλεγμένους δημοσίους υπαλλήλους από τέσσερα κράτη-μέλη για να καταλήξουν επί της μελέτης Εραλίνη και να ε, απαλείψουν τις διστάμενες απόψεις, τις διαφορετικές απόψεις. Ε, επρόκειτο να περιοριστεί η βλάβη που υπέστη η ΕΦΣΑ από όλα αυτά και να πάρει κομισιόν γρήγορα αποτελέσματα και να προστατεύσει τη φήμη αυτών που προστατεύουν τα μεταλλαγμένα εδώ και μία δεκαετία στην Ευρώπη. Άρχισε η δουλειά, ε, και η Κομισιόν ε, επιχείρησε να ε, δυσφημίσει τον καθηγητή Σεραλίνη και τους συνεργάτες τους. Ξέρουμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για αυτή την εκστρατεία που κορυφώθηκε στη δήλωση ε, της ΕΦΣΑ από 28 Νοεμβρίου από πού πήραν την εντολή, με τι δικαίωμα αξιολόγησαν ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση τα, την έρευνα αυτή, ακούστηκαν άλλοι ερευνητές και κρατη Μια μικρή ομάδα προωθήθηκε από το γραφείο τύπου χωρίς διαβουλεύσεις και με πλήρη επίγνωση ότι θα γινόταν δεκτή από κάποια ΜΜΕ, ως, από τα ΜΜΕ που θα έσπευδαν να την αναγνωρίσουν ως ε, επίσημη άποψη της Κομισιόν και της ΕΦΣΑ. Αυτό είναι κατάχρηση εξουσίας και κατηγορώ και την Κομισιόν και την ΕΦΣΑ που τη συνομότησαν για να ε, υπονομεύσουν την αξιοπιστία μιας απόλυτα ακέραιης επιστημονικής ομάδας. Ήταν, είχα και πολλά, ε, ε, πολλές ελλείψεις η απόφαση της ΕΦΣΑ και επί μία δεκαετία ε, δεν ε, ακολούθησε σωστή διαδικασία για τα μεταλλαγμένα ε, σε βάρος της ασφάλειας των καταναλωτών. Η οικογένειά μου και εγώ είχαμε υποθέσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να δώσει προτεραιότητα στη δημόσια υγεία, ενώ φαίνεται ότι η βασική προτεραιότητα που έχει είναι η προστασία μιας διεφθαρμένου, ενός διεφθαρμένου κλάδου μεταλλαγμένων που δεν ωφελεί τους καταναλωτές και θέλει να προστατεύσει τη φήμη των μελών της ΕΦΣΑ και των πάνελ δεν αξίζουν προστασία από κανένα όμως γιατί κατά τη γνώμη μου είναι ένοχοι για συνεχιζόμενη, συνεχή αμέλεια, ε, προκατάληψη, ανεπάρκεια στη δουλειά τους. Ε, ε, πρέπει, πρέπει να εμποδιστούν πριν κάνουν και άλλη ζημιά. Η Επιτροπή Αναφορών τώρα του Κοινοβουλίου τι μπορεί να κάνει. Δεν είμαι βέβαιος. Αλλά εγώ θέλω να αναλυθεί κατεπίγουσα δράση κατά της Κομισιόν και της ΕΦΣΑ που δεν βλέπουν αυτά που βλέπουν οι άλλοι γιατί δεν θέλουν να κοιτάξουν εκεί που πρέπει. Ευχαριστώ. Thank you. Per la Ευχαριστώ εκπρόσωπος Κομισιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έτσι να υπενθυμίσω στον κύριο Τζομπράν ότι η ΕΦΣΑ δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μεροληπτεί υπέρ της βιομηχανίας γιατί πρόκειται για ανεξάρτητο φορέα που έχει αυτή την εξαρτησία από το ότι τα πανελίδια συναπαρτίζονται από ε, άτομα από διαφορετικούς άλλους φορείς. Εξού και η πολυγνωμία και η πληθωρικότητα και γι' αυτό έχουμε την επιλογή λοιπόν των μελών με κάποια διαδικασία πάρα πολύ αυστηρή, προσεκτική οπότε έχουμε και αυτές τις δηλώσεις ε, συμφέροντος ε, οι οποίες χτενίζονται από το προσωπικό της υπηρεσίας και από την ε, Επιτροπή Επιλογής. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι φεύγουν από την ΕΦΣΑ και μετά ξαναγυρίζουν στην βιομηχανία, αλλά, αλλά αυτό δυστυχώς δεν απογορεύεται από τον νόμο. Αυτό ισχύει όταν κάποιος έχει κάποια σύμβαση ορισμένου χρόνου, όταν λήξει αυτή είναι ε, ελεύθεροι να πάνε αν θέλουν στη βιομηχανία, να, να ξαναγυρίσουν σε κάποια κυβερνητική υπηρεσία. Από την άλλη μεριά έχουμε τις κατευθύνες γραμμές τις οποίες χρησιμοποιεί η ΕΦΣΑ ούτως ώστε να είναι η θέση να αξιολογήσει τις ε, αιτήσει ε, ιδιωτικών εταιριών. Οπότε αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ε, είναι πάρα, πολύ λεπτομερείς. Σα παραπέμπω στην δεύτερη αναφορά. Τώρα, σε σχέση με αυτέ τι επικρίσει όσον αφορά την προσβασιμότητα στα έγγραφα, οι αιτήσει καλύπτονται, διέπονται από έναν κανονισμό της Επιτροπής. Και εμείς υποχρεούμεθα να δώσουμε προσβασιμότητα εις ε, πραγματικά περιστατικά, εις επιστημονική τεκμηρίωση, ό,τι ζητείτε και όποτε ζητείτε. Υπάρχουν φυσικά και κάποιο είδου ε, στοιχεία τα οποία είναι εμπιστευτικά, αλλά αυτά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και αυτό γίνεται μόνο όταν αυτά τα στοιχεία είναι εδώ να παραλάσσουν τα εμπορικά συμφέροντα ε, κάποιε εταιρείε. Τώρα, όσον αφορά αυτή την Γεωργιανή, κατά το οποίο αφορά τον κύριο Σεραλίνη, το 613 δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε 8 αιτήματα για πρόσβαση στο έγγραφο και μεταξύ αυτών από τον κύριο Διδόκτρα Σεραλίνη, οπότε και εμείς έχουμε παράσχει όλες τις ζητηθείς πληροφορίες. Μας δεν μπορεί κανείς να πει ότι αποκρύπτουμε τα επιστημονικά δεδομένα από τους ε, ε, αναφέροντες. Τώρα όσον αφορά την ανεξάρτητη έρευνα, όσον αφορά ε, την προσβασιμότητα σε αυτούς τους πόρους, είχε γίνει αυτή η, η, αυτή, ε, αυτό το διάβημα προς τον κύριο Μπράιον και σας υπενθυμίζω απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε μια σειρά προγράμματα ερευνητικά, το οποίο είναι εξάρτητο όσον αφορά την, ε, την, την, την ε, το την αυλαβή αυτά τέλο τα, τα μεταλλαγμένα. Τα δύο τελευταία προγράμματα τα οποία ακόμα τρέχουν είναι το πρόγραμμα GRASS και το GMC Food. Ε, αυτά πέρασαν από εμά και επομένω τα χρήματα αυτά έχουν δοθεί για χρηματοδότηση ανεξαρτήτων μελετών. Επίσης, έχουμε αυτή την περίφημη μελέτη του Δ. Σεραλίνη Όντως, άπως και τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στα ΜΜΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβληματίστηκε με τα αποτελέσματα, αλλά και με τις φωτογραφίες. Είδαμε εκεί αυτούς τους όγκους, τους μεγάλους κλπ. Και, όλος ο κόσμο και εμείς επίσης ε, που τις Και γι' αυτό το λόγο και ζητήσαμε από την ΕΦΣΑ να μας ε, διαβιβάσει ε, σύντομα, όχι όχι σε εξάμεινο, σύντομα, σε δυο τρει εβδομάδες να μας γνωμοδοτήσει όσον αφορά αυτή τη μελέτη. Και έτσι γνωμοδότησε η ΕΦΣΑ ε, επιβεβαιώθηκε με μια δεύτερη γνωμοδότηση την περασμένη εβδομάδα. Οπότε και αυτά όλα συνάδουν προς τη γνωμοδότηση άλλων έξι επιστημονικών φορέων κρατών μελών, αλλά και από άλλους φορείς επιστημονικούς τρίτων χώρων. Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, ΗΠΑ. Οπότε, μια σειρά επιστημόνων επιβεβαίωσαν την άποψη της ΕΦΣΑ. Οπότε και εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια κοινή άποψη από των επιστημόνων. πρεσβεύουν τα ίδια όπως και η ΕΦΣΑ. Όλα αυτά, διότι αυτό το οποίο να ξέρουμε είναι κατά πόσον η ΕΦΣΑ μπορεί να κατηγορηθεί ότι ε, συνομωτεί, ότι τώρα πάντων τα έχει βρει με αυτές τις εταιρείε. Είμαι θα πεπισμένη ότι η ΕΦΣΑ είναι αμερόληπτη και ανεξάρτητη και 100% αρνούμεθα και ακατηρμικά αυτού του είδους τις ε, κατηγορίας συνέργειας. Και για τον Δ. το ίδιο ισχύει. Οπότε, η Γενική Διεύθυνση για την Υγεία και τους Κατάλλωτες έχει ως στόχο την προστασία της υγείας. Αυτό επιβιώνεται από όλες αυτές τις ε, επιθέσεις. Είτε μέσω δικαστηρίου, είτε άμεσες κατηγορίες που διπώνται από τις εταιρείες κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. περισσότερε αυτέ τι περιπτώσει φυσικά κερδίζουμε το δικαστήριο. Όλε αυτέ οι καταγγελίε, είτε για μεταλλαγμένα είτε για φυτοφάρμακα, όλε αυτέ αφορούν καταγορίε των εταιριών ότι είμαστε πολύ αυστηροί. Όμω τελικά δικαιωνόμαστε. Επομένω, απορρίπτουμε τα όσα περιέχει αυτή η αναφορά. Ιδίω σε σχέση με την συνέργεια που φερόμεθα ότι έχουν διαπράξει. Και όσον αφορά την έλλειψη αμεροληψία και εξαρτησία τη ΕΦΣΑ. Και όσον αφορά επίση το ότι δεν ασχοληθήκαμε όσο θα έπρεπε με αυτό το πρόβλημα. Οπότε θεωρούμε ότι ασχοληθήκαμε με όσο γίνεται δυναμισμό. Όσο χρειάζεται, ούτω ώστε να μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε το θέμα αυτή τη έρευνα του κ. Σεραλίνη. Βεβαίω, και ε, προβληματιστήκαμε, αλλά, αλλά το σύνολο της επιστημονική κοινότητα και όχι μόνο η ΕΦΣΑ απεφάνθησαν με τον ίδιο τρόπο. Άρα και εμείς πιστεύουμε ότι οι μελέτες από των οποίων στηρίζονται κατηγορίες δεν είναι και τόσο επιστημονικά αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Κύριο Στάιμπερ. Κύριο Στέιλορ. I do Ζητώ συγγνώμη. Δεν ε, μπορούσα να πιστέψω τα όσα μόλις άκουσα. Αλλά σας ευχαριστώ πολύ, Κομισιόν. Εδώ θέλω να υποστηρίξω και την αναφορά του Brian John, καθώς ε, και την αναφορά 305 που θα συζητηθεί. Η ΕΦΣΑ πρέπει να προβαίνει σε αναλύσει κινδύνου ό,τι αφορά την ασφάλεια τροφίμων και των ζωοτροφών ε, και προβαίνει σε κάποιες συστάσεις και αποφάσει που φύγουν την υγεία εκατομμυρίων πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ε, εγώ καταρχήν ανησυχώ πάρα πολύ όταν ακούω για τις ε, πολλές σφερόμενες ελλείψεις σε σχέση με τα γενετικά τροποποιημένα και επίσης ε, με ανησυχεί το ότι η Κομισιόν ε, απορρίπτει την έκθεση Σιρελίνη με το πολύ γρήγορο συμπέρασμα ότι ήταν ε, κακή η μεθοδολογία Σεραλίνη. Νομίζω ότι αυτό ήταν πάρα πολύ βιαστικό. Όταν, ε, εξετάζ, όταν θεωρήσουμε ότι αυτά τα προϊόντα πολλούνται για τρόφιμα, για ανθρώπινη κατανάλωση και κατανάλωση από το ζωέ, εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό. Δεν νομίζω ότι η αρχή της πρόληψης που ανέφερε ο κύριος Τζον έχει ληφθεί διόντως υπόψη. Και ακόμη και αν έκθεση ρελίνη τόνιζε αρνητικά ε, αντίκτυπο, αρνητικό αντίκτυπο σε ποντίκια μακροπρόθεσμα, η Κομισιόν τι μας είπα, η ΕΦΣΕ είναι ένα εξάρτητο όργανο που μπορείτε να το πιστέψετε αλλά <laughs> φυσικά αν το λέει η ΕΦΣΑ αυτό, δεν θα ε, λέει κάτι διαφορετικό, έτσι. Αν ε, λοιπόν είναι μεροληπτούσαν, αν ε, τελικά κάλυπταν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα, αυτό ακριβώς θα έλεγαν. Και αυτό παρά το ότι πολλοί ανεξάρτητοι επιστήμονες, αμερόληπτοι επιστήμονες, ε, υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή στην οποία υποστηρίζουν τη μεθοδολογία Σρελίνο. Επομένω δεν ξέρω πού πάμε από εδώ και πέρα, γιατί φαίνεται ότι έχουμε την ΕΦΣΑ. Ακούσαμε ε, ότι θεωρείται μεροληπτική, ακούσαμε την Κομισιόν να μα λέει «Μα όχι, η ΕΦΣΑ ξέρει γιατί πράγμα μιλάει» και μιλάμε και για ένα καταναλωτή που βρίσκεται σε κίνδυνο και θέλω να ακούσω κάτι ένα συγκεκριμένο τρόπο να προχωρήσουμε προς τα μπρος. Ίσως μήπως ε, να δούμε αυτό το πάνελ γαματάφ όμικρον και να αντικαταστήσουμε τα μέλη του με κάποιους που δεν έχουν προσωπικό συμφέρον από τη βιομηχανία γενετικά τροποποιημένων. Δεν νομίζω ότι είναι και πολλά να ζητάμε από ένα φορέα που ασχολείται με την ασφάλεια των τροφίμων μας. Έτσι λοιπόν ε, θέλω να απευθυνθώ στον νέο Επίτροπο Σάνκο να απαιτήσει από τις εταιρείες να κάνουν μακροπρόθεσμες δοκιμές σε όλα τα προϊόντα. Αυτή η ρουρέι τον οποίο είδατε φωτογραφίες, δεν είναι ατύχημα. Είναι, δεν είναι κάτι που απλώς τυχαία έγινε, έγινε υπό συγκεκριμένες δοκιμές. Και Πραγματικά με που η Κομισιόν με τόσο γρήγορο τρόπο τα απορρίπτει όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Γκαρσές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην έκθεση του 2010 σε μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που εστάλει στην Επιτροπή Αναφορών. Η Επιτροπή έλεγε, η Κομισιόν έλεγε ότι θεωρούσε την προστασία της υγείας, της ανθρώπινης υγείας και των ζώων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και δεσμεύεται στο να εγγυθεί ότι οι σπόροι, τα τρόφιμα και οι γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές θα ε, δοθεί άδεια σε αυτά μόνο όταν δεν επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, ούτε για το περιβάλλον. Λοιπόν, αυτή τη δήλωση πρέπει να την υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον κύριο προσανατολισμό των εργασιών σε σχέση με τις επιπτώσεις των καμεταφόμικρων στην ανθρώπινη υγεία. Επομένως, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι επιβάλλεται για μια ακόμη φορά η απέτηση, αυτή η αρχή της πρόληψης να ληφθεί υπόψη και να μην απομακρυνθούμε και καταλάβουμε εντάχει θέσεις μπροστά σε τόσο σημαντικά γεγονότα όπως αυτά που καταγγέλει η έκθεση. Αναφεσβητητά, το είπε εδώ και η Κομισιόν προλίγου. Βρισκόμαστε εδώ σε μια στιγμή όπου συγκρούνται πολύ ισχυρά συμφέροντα κάθε είδους και δεν είναι η πρόθεσή μου εδώ να την αλύσω βεβαίως. Αλλά αναμφισβήτητα αυτή η σύγκρουση συμφερόντων γίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά και σε άλλες ε, περιπτώσεις. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σόφρονες πριν να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα, γνωρίζοντας ότι η επιστημονική κοινότητα έχει αποκλίνουσες απόψεις. Υπάρχουν αιτιολογημένες επιστημονικά απόψεις που μας οδηγούν σε αποκλίνοντα συμπεράσματα. Σε αυτόν τον βαθμό, εγώ νομίζω ότι πρέπει να απαιτήσουμε από την εύσα να είναι και αυτή σόφρον και να μην βιαστεί στην λήψη αποφάσεων. Ίσως θα ήταν απαραίτητο να συνεχίσουμε να ζητάμε περισσότερες εκθέσεις και να συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιστημονική Κοινότητα κυρίως στην ακαδημαϊκή επιστημονική κοινότητα, που δεν σχετίζεται ούτε άμεσα ούτε έμεσα με τομεακά συμφέροντα. Γι' αυτό από αυτή τη διτή θέση, δηλαδή της αρχής της, προ... της πρόληψης και της οφροσύνης, θα έπρεπε να θεωρήσουμε ότι παραμένει ανοιχτό αυτό το θέμα, ότι θα συνεχίσουμε να το διαρευνούμε και ότι η έκθεση της ΕΦΣΑ που έχουμε στο φακελό μας δεν θεωρηθεί ως μια οριστική θέση, μας μια έσχατη θέση. Όταν θα προσανατολίσει τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το αντίθετο, να θεωρηθεί ότι αυτό το θέμα χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, περαιτέρω μελέτη και η αρχή της πρόληψης θα πρέπει να εφαρμόζεται εδώ. Και ίσως θα άξιζε τον κόπο να δούμε τι, πώς, το πόσο είναι εφικτό να καλέσουμε τον καθηγητή Σερελίνη να έρθει εδώ και να μας παρουσιάσει την έρευνα που υλοποιήθηκε και να μπορέσουμε και εμείς με τα ίδια μας τα αυτιά και τα μάτια να διαπιστώσουμε κατά πόσο είναι αληθή τα όσα λέγονται. Okay. Σύντομα, δύο λόγια για την Κομισιόν σχετικά με την ανικανότητα. Δεν είναι ότι δεν είναι εντάξει και σωστοί οι άνθρωποι. Ένα, πρέπει να δουλέψουμε με αντικειμενικά κριτήρια, όπως ότι θα είναι ελεύθερη από σύγκρουση συμφερόντων. Και όταν είναι κανείς τόσο κοντά στο κλάδο της βιομηχανίας, όπως είναι αρκετά μέλη της ΕΦΣΑ, γιατί παλιά ήταν πριν στη βιομηχανία, κάποιοι επανέρχονται στη βιομηχανία. Και όταν δείτε αυτό τον κλάδο της βιομηχανίας, βλέπω ένα μεγάλο δίκτυο που στο κέντρο κάθε τη Μονσάντο και βλέπετε πώς καλύπτουν τόσα συμφέροντα σε όλη την Ευρώπη. Μεγάλες διεθνείς εταιρείες που είναι ε, μικρά πλοκαμάκια της Μονσάντο. Ε, πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η Μονσάντο αρνείται ότι κατασκευάζει τερατώδη εισιτήρα που δεν καταπολεμούνται με τα... που δεν καλύπτονται με τα συνήθης ζανιοκτώνα και ότι τώρα πέφτει η, η, η ανθεκτικότητα αυτών των ε, καλλιεργειών τα βλέπουμε και φέτος κάνουν πάλι τα ίδια. Άρα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η Κομισιόν. Δεν μπορεί να λέει και να δηλώνει ότι η ΕΦΣΑ είναι ανεξάρτητη. Βεβαίως πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Αντικειμενικά όμως δεν είναι. Αυτό είναι βέβαιο. ή όταν πρόκειται για κλινικές μελέτες κλπ. Όλο λέμε δεν τα ξέρουμε, ενώ υπάρχουν, τα ξέρουμε. Πώς θα τα εντοπίσουμε. Ας κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή, ας σταθούμε κοντά στους αναφέροντες και να πούμε Εμείς είμαστε εδώ για τους πολίτες και νομοθετούμε για τους πολίτες. Οι πολίτες μας καλούν να τους προστατεύσουμε. Εμείς είμαστε η Επιτροπή των Πολιτών. Και αν λείπει διαφάνεια, που λείπει σε αυτούς τους οργανισμούς, και η ΕΦΣΑ είναι από τους πιο σημαντικούς, είχαμε και με την έμα μεγάλους καυγάδες. Δεν ξέρω αν ο οργανισμός αίμα είναι ακόμα λειτουργεί έτσι όπως πριν και δίνει εγκρίσει σε προϊόντα πως είναι ένα για την, ε, το θερμιφλού που είναι για την πανόλη των χείρων. Θέλει μεγάλη προσοχή σε όλα αυτά. Δεν, δεν μου άρεσε που είπατε ότι είναι καλοί άνθρωποι αυτοί και δεν ε, είναι ανεξάρτητοι και δεν έχουν συμφέροντα και ότι αυτούς βρήκαμε, αυτή είναι η καλύτερη που θα μπορούσαμε να βρούμε, ενώ αυτοί επηρεάζονται από τη βιομηχανία. Ευχαριστώ κύριο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι εύκολο για την ΕΦΣΑ ούτε για την Κομισιόν να είναι αντικειμενική. Πάντως κάνει εντύπωση ότι η ΕΦΣΑ δεν εξαιρείται από την κριτική. Δηλαδή είναι άκομψη η χειρισμή της και νομίζω ότι ήρθε η ώρα και η διοίκηση και ο νέος Επίτροπος Υγείας και Κομισιόν να δουν το θέμα αυτό και να βάλουν σαφείς κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων. Εγώ δεν είμαι τόσο ακραίος όπως η συνάδελφος Άουκεν που λέει ότι Κανένας από τη βιομηχανία δεν πρέπει να συμμετέχει εκεί, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να ε, έχουμε διαφανείς, ξεκάθαρους κανόνες και να μην γίνονται τέτοιες άκομψες κινήσεις ε, όπως του κυρίου Κρούεν, ο οποίος είχε πολλά συμφέροντα σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Ίσως έχουμε έτσι μια ευκαιρία να ε, αντιμετωπίσουμε τη δημόσια κριτική γιατί τα θέματα αυτά είναι πράγματι πολύ αμφιλεγόμενα. Πολλοί συνάδελφοι από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, συμφωνούν μαζί μου και λένε ότι φτιά, ε, ε, παρουσιάστε σαφείς κανόνες, βάλτε την ΕΦΣΑ να τους ακολουθεί και την αίμα και την ΕΦΣΑ και όλους ούτως ώστε να ησυχάσουν τα πνεύματα. Γιατί σε κάθε απόφαση είναι επώδυνο ότι ξεσπούν φασαρίες μετά από κάθε απόφαση. Αυτό βλάπτει και το κύρος της ΕΦΣΑ και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερον, πρέπει να πούμε ότι ήταν λίγο περίεργο με τη μελέτη Σεραλίνη. Εγώ δεν είμαι επιστήμονα, αλλά είναι περίεργο πόσο γρήγορα ε, αντέδρασε η Κομισιόν με προκατάληψη. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μπουν σε περισσότερες λεπτομέρειες, να κοιτάξουν ποια θέματα ήταν ε, που ε, επιδέχονταν κριτική και θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν αυτά τα βασικά σημεία κριτικής που λέτε ότι τα συμμερίζονται πολύ να μας τα δείξετε και μας για να καταλάβουμε πού έκανε λάθος κατά τη γνώμη σας η έρευνα γιατί εγώ πήρα πληροφορίες, το είπαν κι άλλοι, ότι αυτά με τις εγκρίσεις ε, των μεταλλαγμένων, αυτό το, ε, η επίδραση, η μακροπρόθεσμη, δεν λήφθη υπόψη επαρκώς. Και το ενδεχόμενο να τα μεταλλαγμένα να επηρεάσουν το κλίμα, του οικοτόπου, τα βιβλιοσυστήματα. Δεν ε, εξετάστηκαν καλά. Εδώ έχουμε μία τεχνολογία που έχει μεγάλο αντίχτυπο στο περιβάλλον και την υγεία μας από ό,τι φαίνεται. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και γι' αυτό η συνθήκη ε, αναφέρει ρητά την αρχή της προφύλαξης. Αν υπάρχουν αμφιβολίες, πάντα θα δράσουμε υπέρ της ανθρώπινης υγείας και υπέρ του περιβάλλοντος. Α, όταν λαμβάνεται μία απόφαση πρέπει να είναι υπεράνω πάσης αμφιβολίας. Δύσκολο, αλλά επειδή εδώ έχουμε αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών που τα απορρίπτουν όλα αυτά και διχάζονται τα κράτη-μέλη, κάποια στιγμή και η Κομισιόν θα πρέπει να αρχίσει να βαράει το καμπανάκι. Γιατί δεν ε, αποδεικνύονται όλα αυτά επιστημονικά και είναι δύσκολο να προχωρήσουμε έτσι. Ε, ε, υπάρχουν ορατόρια, κανείς δεν τηρεί τους κανόνες, άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση δυσάρεστη για όλους, και για τα κράτη και για τους πολίτες και για σας. Καλό είναι λοιπόν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε ε, και την κριτική στην ΕΦΣΑ. Τώρα, ε, για το οικονομικό όφελος από αυτή την τεχνολογία, γιατί μας λένε ότι αυτή θα σώσει την ευρωπαϊκή γεωργία, πράγμα που εγώ το αμφισβητώ. Ίσως όμως μπορούμε να πούμε δύο λόγια και πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ξέρουμε ότι αυτή η τεχνολογία προχωράει ε, σε διαφορετικό βαθμό στα διάφορα κράτη-μέλη. Να δούμε τι κάνουν στη γεωργία σε εθνικό επίπεδο καθένας. Ε, καλό είναι να παραμείνει λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους ανοιχτή η αναφορά και να συνεχιστεί η συζήτηση στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μιράντα. Ευχαριστώ πρόεδρε πέρα από το αυτό το θέμα είναι δημοσίου συμφέροντος για πολλούς από εμά πρόκειται και ένα θέμα υπεράσπισης των δικαιωμάτων ε, των, ε, ε, του εκλογικού μας σώματος, των γεωργών, των πολιτών που ζητούν πληροφορίες για τα γενετικά τροποποιημένα. Εγώ μιλάω για την περίπτωση της πατάτας. Προέρχομαι από μια χώρα που παράγει πατάτα, μία από τους κύριους παραγωγής πατάτα στην Ευρώπη, όπου είδαμε σε διάφορες ζώνες ε, γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες ε, και είναι τόσο κοντά αυτές οι καλλιέργειες η μία στην άλλη και δεν υπάρχει εγγύηση για το που είναι γενετικά τροποποιημένες παραγωγές και ότι είναι διαχωρισμένες από την ε, κανονική παραγωγή της πατάτας. Όμως τελικά πώς θα εγγυθούμε την ομοθεσία, πώς θα εγγυθούμε ότι οι παραδοσικές καλλιέργειες συνυπάρχουν με τις γενετικά τροποποιημένες και η περίπτωση της επιμόλυνσης, στην περίπτωση του μελιού. Η ίδια η ουσία των φυτών δεν μένει, ξέρετε, γύρι στατική, δεν υπάρχουν σύνορα, ε, υπάρχουν μεταφορά, υπάρχει μεταφορά των καλλιεργιών από τη μία στην άλλη, γιατί δεν είναι σε επαρκή απόσταση και Θέλω να αναφέρω ε, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 6ης ε, Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την οποία ε, χρειάζεται συγκεκριμένη διαδικασία για την μελισσοκομεία όταν βρίσκονται κοντά γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες. Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες χωρίς καν να γίνονται κάποιοι έλεγχοι ή πειράματα όπως έγινε στην Γαλλικία ή το γεγονός ότι βλέπουμε αυτό το άνοιγμα προς την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε μια νέα ποικιλία πατάτας ε, που γεννείται από μετάλλαξη ενώ έχουμε ε, φυσικές ποικιλίε ε, και πατάτες που τις καλλιεργούμε για την κατανάλωση από το ζωή. Εμείς τι θέλουμε, μια βιώσιμη γεωργία ή μια γεωργία όπου τελικά θα προωθεί καλλιέργειες που έχουν συνέπειες αρνητικές σημαντικές για τον άνθρωπο και για τα ζώα. Και τέλος θέλω να κάνω μία αναφορά σε ένα ζήτημα που μου φαίνεται σημαντικό και είναι η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων ε, καθώς υπάρχουν επιστημονικές αμφιβολίες σε σχέση με το πόσο επικίνδυνο είναι για την, την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον. Αναφέρθηκε εδώ από αρκετού συναδέλφους το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό, ο αναφέρον έχει το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ από όσο απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρε, αποκόμισε την εντύπωση ότι έχει υιοθετήσει παθητικό ρόλο και επαναλαμβάνει αενάως Ξέρουμε τι κάνουμε. Ξέρουμε ότι ξέρει η αίθουσα τι κάνει. Είναι υπεύθυνοι επιστήμονε. Είναι ικανότατοι. Γιατί να του αμφισβητούμε. Λυπάμαι. Φοβάμαι ότι αμφισβητείται εντόνω η αίθουσα από πάρα πολλού αμερόληπτου, ανεξαρτήτου επιστήμονε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε αναλυθεί ισχυρισμού σε σχέση με το, το, το δίθεν αντίκτυπο, τη δίθεν υποδοχή των εκθέσεων της ΕΦΣΑ. Είναι Καναδά, είπα Νέα Ζηλανδία. Φυσικά αυτοί αυτοί έχουν τόσα συμφέροντα, Τετοιε πολιτικέ έχουν υπέρ των μεταλλαγμένων, γιατί επίσης ε, υπάρχει και άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι άλλοι επιστήμονε. πρόκειται για του επιστήμονε του ανεξαρτητού, οι οποίοι δεν έχουν συμφέροντα, δεν, δεν, δεν έχουν ανάμεση με τη Μονσάμι, με τις αριστερίε. Και ε, στη μελέτη εκείνου του καθηγητού ε, οι απόψεις τους και επομένω γι' αυτό και εμεί θέλουμε το, το, το κοινοβούλιο μα βοηθήσει σε αυτήν την προβληματική πρόεδρο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλου που συμμετείχαν στη συζήτηση. Σίγουρα δεν κλείνει το ζήτημα εδώ, γιατί και απάντηση τη Κομισιόν σε σχέση με την αξιολόγηση τη συμπεριφορά ε, τη ΕΦΣΑ, τη τάση τη ΕΦΣΑ και στι νομοδοτήσει που εκφράζει, δεν έχει ικανοποιήσει όλου του συνάδελφου που θεωρούν ε, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αξιολογούμε το ζήτημα. Εγώ νομίζω ότι ε, κατόπιν πρόταση του κ. Γκαρτσέ, νομίζω ότι μπορώ να δεκτό και την πρόταση να συναντήσουμε το συντάκτη της έκθεσης. Θα μπορούσε να είναι κάτι ενδιαφέρον για να δούμε επί της ουσίας κάποια ζητήματα και να μπορέσουμε να κρίνουμε και καλύτερα και τη θέση της Κομισιόν που υποστηρίζει απόλυτα τις εργασίες και τις δραστηριότητες της ΕΦΣΑ. Αν συμφωνείτε λοιπόν θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και θα καλέσω και τον υπεύθυνο της έκθεσης, ε, αλλά και τους επιστημονιστές για να μπορέσουμε να ε, δούμε ερετέρω εις βάθος το ζήτημα αυτό. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ωραία. Επομένως, σας περάσουμε στις δύο επόμενες αναφορές. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναδέσω το λόγο στον κύριο Μπρέιαν Τζον, όμως σας ζητώ να είστε πιο σύντομος ε, για να επανέλθουμε στο θέμα με μια διαφορετική οπτική. Δύο λεπτά σας δίνω για να παρουσιάσετε τη θέση σας για αυτό το τελευταίο τμήμα που ε, ουσιαστικά σχετίζεται και με την αναφορά 305 του 2010. Thank you, Chair. Um, I'll try to... Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν τη γραπτή παρουσίαση και υπάρχουν περισσότερε λεπτομέρειες εκεί. Εκ μέρου ε, των επιστημόνων που έστειλαν ε, το 2010 αυτή την επίσημη, αυτό το επίσημο εγγραφό και όσοι το υποστηρίξαν, ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και πάλι το ότι ε, ο κανονισμός είχε ε, ως στόχο να θα εφαρμοστούν οι κανόνε που διέπουν την έγκριση των γενετικών τροποποιημένων ε, τροφίμων. Εμεί πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κοινοβουλευτικό έλεγχο ε, και στο ιστορικό τη ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ έγιναν μυστικέ διεργασίε. Είμαστε αντίθετοι στο ρόλο που έπαιξε η ΕΦΣΑ στην κατάρτιση αυτού του κανονισμού και θεωρούμε ότι η ΕΦΣΑ τώρα διαδραματίζει ένα παράνομο ρόλο στην ε, χάραξη τη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, στους ΓΔ Η ΕΦΣΑ έχει πολύ μεγάλη ευχαίρεια που θα την ασκήσει στο μέλλον στην διαδικασία ανάλυση όταν αυτή η ευχέρεια γράφεται στο νόμο και ασκείται κατόπιν από την ΕΦΣΑ, ε, η οποία είναι μεροληπτική απέναντι στη βιομηχανία και θεωρεί τους γάματα φόμικρον τότε έχουν δικαίωμα αντίρρησης οι πολίτες της Ευρώπης. Έχουμε αρκετά κυρία σημεία. Η ΕΦΣΑ εξακολουθεί να βλέπει συγκριτικέ ε, μελέτε κινδύνου ω μια πρότυπη διαδικασία, όπω ε, δέχεται και την ε, ουσιαστική ισοδυναμία και την έννοια του γενικά ασφαλού. Υπάρχουν κανονισμοί για τα γενετικά τροποποιημένα που ουσιαστικά μπορούν να προκαλέσουν αλλεργία ή τοξικότητα. Έχουμε νέε χημικέ ενώσει που δεν μπορούν να ευρεθούν ε, όταν χρησιμοποιούνται δοκιμέ για τι γνωστέ ουσίε και θεωρείται έτσι ότι το φυτό είναι ασφαλό να καταναλωθεί. Και η ΕΦΣΑ και η Κομισιόν έχουν εγκαταλείψει τώρα την αρχή τη πρόληψη, από όσο βλέπω ε, παρά τα όσα προβλέπει η οδηγία και αυτό ο εφαρμοστικό κανονισμό, τον οποίο μιλάμε δεν αποτεί να γίνουν δοκιμέ σε σχέση με την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον ε, που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των γάματα μικρών και δεν ακολουθείται μία σταδιακή διαδικασία. Σύμφωνα με τον κανονισμό και η βιομηχανία και οι νομοθέτες μπορούν να απορρίψουν σημαντικές αλλαγέ, είτε ε, στα φυτά είτε ε, στα ζώα χωρίς να τα θεωρήσουν σχετικά και χωρί να ορίσουν αυτό τι σημαίνει. Παρόλο που οι 90 ημέρες δοκιμών είναι τώρα υποχρεωτικέ η ΕΦΣΑ θεωρεί ε, ότι μπορεί να μην δέχεται αυτές τις μελέτες όταν το θεωρεί κατάλληλο. Πρέπει να μην έχουμε ισογενικές γραμμές συγγενικές και... Συγγνώμη, μπορείτε να ολοκληρώσετε, λέει η Πρόεδρος. Έχω και κάποια άλλα σημεία, αλλά θα φτάσω στο συμπερασμά μου, αν ε, θέλετε να τα συζητήσετε αυτά. Λοιπόν, η διαδικασία αξιολόγηση ε, κινδύνων ε, ουσιαστικά γίνεται με ταχεία διαδικασία και θα υποσκάψει το σημερινό κανονισμό και επίσης θα ληφθούν αποφάσεις κατά του Συμβουλίου Περιβάλλοντος που ζητούσε μεταρρύθμιση. Ενώ ο εφαρμοστικό κοσμισμό στη σημερινή του κατάσταση θα οδηγήσει σε εγκρίσει ε, επικίνδυνων γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών που θα έχουν αρνητικέ συνέπειε. Επίση, θα συμπεριλάβει μια σειρά παράνομων πολιτικών αλλαγών. Ζητάμε από το Κοινοβούλιο να απορρίψει τον εφαρμοστικό κανονισμό και να λάβει βήματα να διασφαλίσει ότι η ΓΔΣΑΚΟ δεν θα ε, το εγκρίνει και το πάνελ της ΕΦΣΑ δεν είναι καθόλου κατάλληλο. Εμείς ε, καλούμε την άμεση διάλυση αυτού του πάνελ και να αντικατασταθεί από ένα οργανό του οποίου τα μέλη δεν έχουν προσωπικό συμφέρον στην ε, βιομηχανία των γενετικά τροποποιημένων και ε, θα προστατεύσουν την υγεία και θα τη βάλουν πάνω από την πολιτική αποτελεσματικότητα. Εκπροσωπώ και άλλους συναδέλφους από όλα μέρη της Ευρώπης και ζητώ να εξεταστεί προσωπικά τα θέματα που έθεσα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πιντέλη και πάλι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στα στοιχεία τα οποία εξετάζονται όσον αφορά αυτές τις περίφημες καθεντήριες της ΕΦΣΑ και την έλλειψη διαφωνία της όλης διαδικασίας. Είχαμε μια σειρά διαβουλεύσεων από ΕΦΣΑ, από Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά αυτές τις νέες καθεντήριες. Ακριβώς όπως λέει και αυτό το είχαμε και διαδικασίες πάρα πολύ διαφανείς, ε, είχαμε όλους τους εμπλεκομένους, όλες τις μη κυβερνικές οργανώσεις που μπορούσαν να τοποθετηθούν και το Κοινοβούλιο επίσης πλάκι, διότι είχαμε ένα σωρό συνομιλίες, επαφές, επιστολή, ε, ανταλλαγή επιστολών με τον ε, πίτρο Φοντάλη, απήντησε εκείνο και το Κοινοβούλιο επίσης πέρασε αυτή την διαβούλευση κατά την φάση της ε, έγκρισης γιατί ακόμα τώρα είμαστε σε φάση της περίσκεψης, της μελέτης γιατί είπαμε ότι πάγωσαν οι πάγωση των διαδικασιών όσο μελετούσαμε την έκθεση Σεραλίνη γιατί θέλαμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα σε αυτό το πρόβλημα της τοξικότητος της μέσοπρόθεσμης. Ε, είναι άκρο αληθές να λέμε ότι αυτό ήταν εκείνη κίνηση, διάβημα ε, το τον ΗΠΑ διότι, διότι από ό,τι γνωρίζω η η Βραζιλία, η Αργεντινή, ο Καναδάς ε, όλοι έκαναν διαδήματα τόσο ώστε να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια τους για τι καθεντήρες γραμμέ. Σαφώς τάξαν κατά τη τοποθέτηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. επιστημονικά την προσέβαλαν. Γιατί αυτό το οποίο θέλαμε στις γραμμέ είναι να έχουμε ε, αυτές τις μελέτες μέσα σε... Είναι, ζήτησε ένα τρίμηνάκι γιατί είπαμε ότι δεν θα... Ε, ε, είπαμε ότι θα πρέπει αυτές οι να προχωρήσουν γιατί το ζήτησαν μη κυβερνικές οργανώσεις. Αν δεν είναι, είμαστε αρκετά αυστηροί έναντι των αναφερόντων. Επίσης, ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να καταλήξουμε την έγκρισή της. Περιμένουμε την άντληση των πλήρων συμπερασμάτων επί της μελέτης ε, σε Ραλίνη, σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιο αλλαγή. Το τον είναι πάντως ότι κάποια στιγμή θα ξανασυντηθεί το θέμα. Αυτά κατά κάποιο τρόπο τηλεγραφικά που θέλαμε να αναφέρουμε η κυρία Πρόεδρε για την υπόθεση. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά κάποιο το λόγο. Από την παρέμβαση τη Κομισιόν μου φαίνεται ότι πρέπει να διατηρήσουμε και αυτή την αναφορά ανοιχτή για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε από κοινού το πόσο επιτυχής ήταν η διαδικασία. Επομένως αφήνουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά για να τη συζητήσουμε σε ένα μετέπειτα στάδιο από κοινού και με την άλλη αναφορά ελπίζω και παρουσία του αναφέροντος ή της αναφέρουσας. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνουμε εδώ αυτό το μπλοκ αναφορών. Ευχαριστώ τον κύριο Brian Τζον, τον, τον αναφέροντα που μας έθεσε αυτό το θέμα και να περάσω στο επόμενο σημείο της ημερής διάταξης. Έχουμε τρεις αναφορές που θα τις δούμε από κοινού. Την 1278, τη 1302 και τη 1525. Και οι τρεις ε, είναι του 2010 και έχουν ως αντικείμενο την φερόμενη παραβίαση ε, των από την Ιταλία της Οδηγίας για την Ανέωση Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου. Είναι ε, παρόντες εδώ δύο από τους αναφέροντες. Θα ξεκινήσω με την πρώτη. Έχουμε την κυρία Πιτσάρτα που θα της δώσω το λόγο για 1,5 λεπτό. Καλησπέρα σας. Εγώ άρχισα να εργάζομαι ως διοικητική βοηθός ε, το κάτι με το 2000-2001 με, ε, ως αναπληρώτρια και το 2003-2004 με καθήκοντα που ανέθεσε το Υπουργείο ε, Παιδείας ε, και η Ιταλική κυβέρνηση Παραβίασε, όσο προβλεπόνται από την 1970 του Ιουνίου του 1999 σύμφωνα με το πλαίσιο σε Unity και σε σχέση με τον ε, εργασία ορισμένου χρόνου ε, σύμφωνα με ε, το διάταγμα 368-2001 και σύμφωνα με το διάταγμα 91-2004 Συγγνώμη, πρέπει να διαβάσετε πιο αργά. Βλέπει λοιπόν ε, ότι ε, όσοι βρίσκονται στη μόνιμη κλίμακα βαθολογίας ε, οι υποψήφοι αυτοί προσλαμβάνονται με σύμβαση αορίστου χρόνου για θέσεις με τον ίδιο σκοπό και σύμφωνα με την ομοθεσία που ισχύει τη στιγμή της πρόληψης όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Εγώ ε, μπόρεσα ε, να αποκτήσω το δικαίωμα στη μετατροπή της σύμβασής μου ορισμένου χρόνου ε, μετά από το πέρας των 36 μηνών ε, της σχέσης εργασίας μου το Υπουργείο ε, για χρόνια καταχράστηκε την εργασία μου μέσω της ε, ανανέωσης σε συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Παρ' όλα αυτά με απόλυσε χωρίς καμία προστασία για το μέλλον. Αυτή η κατάσταση καθορίστηκε από ε, περικοπές το 2008 στο 2011 και επιδεινώθηκε και από άλλες διατάξεις που θετήθηκαν από το Υπουργείο όπως ήταν το διάταγμα του 2010 και είχε να κάνει με την επαγγελματική κινητικότητα των σχολικών συνεργατών και το διάταγμα 17-2011 σε σχέση με την κατάργηση της επαγγελματικής κινητικότητας και τα δύο νομοθετήματα αφαίρεσαν το 40% των εισόδων σε σχέση με τους ε, διοικητικούς υπαλλήλους Έχουμε επίσης το νόμο 111-2011 ε, σε σχέση με την, την ακούσιο πέρασμα ε, των ακατάλληλων εκπαιδευτικών ε, στις κενές θέσεις και το νόμο 95-2012 σε σχέση με τους μη κατάλληλους εκπαιδευτικούς που περνούν για να καλύψουν τις κατάλληλες θέσεις. Επίσης το Υπουργείο για πολλά χρόνια μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την εργασία μου ε, υιοθετώντα μια διακριτική συμπεριφορά. Βάσει της ανανέωσης των συμβάσεων ε, με οδήγησε στον εξαρτώμαι οικονομικά μόνο από αυτή την απασχόληση ε, και ουσιαστικά δεν είχα καμία άλλη εναλλακτική προοπτική εργασίας. Επομένω, δεν μπορώ πλέον να εγγυθώ στην οικογένειά μου τα απαραίτητα προς το ζήν και αυτό με βάζει σε ένα μεγάλο, ε, ένα μεγάλο αγχός και υπάρχουν επιπτώσεις στην ε, ψυχική και σωματική μου υγεία. Πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο η Ιταλία να εφαρμόζει τις ε, την κοινωτική νομοθεσία που επιβάλλει καθήκοντα, ενώ αντίθετα όταν προβλέπονται κάποιες διατάξεις πιο ευνοϊκές σε σχέση με την εθνική νομοθεσία να θεωρεί ότι η κοινική νομοθεσία δεν είναι δεσμευτική, αλλά απλά δίνει προσανατολισμό. Ε, έτσι λοιπόν, όταν ε, μόνο τη συμφέρει την Ιταλία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να με βοηθήσει να ε, μπορέσω να αποκτήσω δικαιοσύνη απέναντι στην παραβίαση των ε, θεμελιωδών μου δικαιωμάτων και ε, ουσιαστικά να οδηγήσει στην άσκηση ε, της διαφύλαξης των δικαιωμάτων μου και να μου δοθεί και η απαραίτητη αποζημίωση. Η Ιταλία συνεχίζει να ασκεί ε, οποιαδήποτε παραβίαση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων που προβλέπονται και στο Ιταλικό Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση με αλαζονία χωρίς να αναγνωρίζει τα αποτελέσματα που προβλέπονται από το Εθνικό Δίκαιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Πατάνη Κιάρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ εκπροσωπώ την κυρία Βαλέρια Πιτσάτη και ε, η πελάτη μου έχει ε, ουσιαστικά για έξι χρόνια προσληφθεί με συμβάσεις ε, ορισμένου χρόνου από το Υπουργείο Παιδείας ε, και την προσλάμβανε από την 1η Σεπτεμβρίου και έλεγαν οι συμβάσεις ε, στις 31 Αυγούστου. Έτσι λοιπόν συνεχιζόταν ε, η εργασία για 6 χρόνια και στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Παιδείας παραβίασε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 70 του 2009 σε σχέση με τον ορισμένο χρόνο εργασίας αλλά και την νομοθεσία που αναφέρθηκε η κυρία, η Πισάρδη. Οι διάφορες συμβάσεις που συνάπτονταν από χρόνο σε χρόνο είχαν την ίδια σχέση εργασίας και είχαν ως στόχο να καλυφθεί η ανάγκη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας στην Κατάνια. Επίσης πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πρόσφατα η κυβέρνηση Μπερλουσκόνη και η κυβέρνηση Μόντι ουσιαστικά πιέζησαν σε ε, μία αναθεώρηση στα ε, συνθήκες που ισχύουν στις προσλήψεις στα δημόσια σχολεία και έτσι ε, από τους σχολικούς συνεργάτες έκαναν τα άτομα αυτά ε, διοικητικούς βοηθούς και μείωσαν ε, ε, και ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί τώρα απασχολούνταν υπό το προφίλ ε, του διοικητικού βοηθού. ουσιαστικά βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη παραβίαση γιατί χωρίς καμία αιτιολόγηση υπάρχει παρέκκληση από την αρχή του δημόσιου διαγωνισμού που προβλέπεται από το άρθρο 97.3 του Συντάγματος. Το Συνταγματικό Δικαστήριο επανέλαβε ότι αυτή η αρχή είναι δυνατό να παρακαφθεί μόνο στην περίπτωση που αυτή η παρέκκληση απαντά σε κριτήρια εξορθολογισμού ή στο να προστατεύσει συνταγματικές αρχές. Στην περίπτωση που εξετάζουμε δεν υπάρχει υπάρχει κανένας λόγος που να αλλαγή, τη διαδικασία ε, αυτή καθώς ε, οι σχολικοί συνεργάτες που συμμετείχαν σε αυτές τις διαδικασίες κινητικότητας ε, ούτε καν έχουν τα απαραίτητα κριτήρια που ζητούνται ε, προκειμένου να μπουν σε μια διαδικασία οριζόντιας κινητικότητας. Έτσι λοιπόν παραβιάζεται το νομοθετικό διάταγμα 165 του 2001 που προβλέπεται ο διαχωρισμός ενός μέρου τους ε, θέσεων που μπήκαν ε, στο διαγωνισμό πάνω του 50%. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η δικηγόρος Δηματέα ε, ζήτησε την άμεση αναστολή των συνεπειών του διατάγματος όμως το δικαστήριο δεν το δέχτηκε και είπε ότι αυτή η διαδικασία της οριζόντιας μετακίνησης δεν πρέπει να θεωρηθεί δημόσιος διαγωνισμός και ε, παρά τις διάφορες αποφάσεις του κυριωτικού δικαστηρίου που καθορίζουν τις διαδικασίες οριζόντιας κινητικότητας ε, ε, ω πραγματικά δημόσιου διαγωνισμού. Συμπερασματικά πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η κατάσταση τη κυρία Πιτσάτη είναι απλώ ε, ένα παράδειγμα γιατί έχει ε, έχουν θυγεί και από αυτή την οριζόντια ε, κινητικότητα αλλά και από τη συνεχή ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου για πάνω από 36 μήνε και άλλοι πολίτε που και αυτοί έχουν παρουσιάσει την ίδια αναφορά αναφορά στην Επιτροπή αυτή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τιμ Ρέντροπ από την Κομισιόν. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι τιμή μου να ενημερώσω τα αξιότιμα μέλη ότι η Κομισιόν άρχισε διαδικασία επιπαραβάση κατά της Ιταλίας πάνω σε αυτό το θέμα Τώρα είμαστε στο, στη φάση της πρόσθετης επιστολής επίσημης κοινοειδοποίησης και περιμένουμε απάντηση από τις Ιταλικές αρχές. Η επιστολή ε, δημοσιεύτηκε 25 Οκτωβρίου φέτος. Είναι πρόσθετη επιστολή επίσημης ε, ειδοποίησης γιατί μετά την αρχική η απάντηση από τις Ιταλικές αρχές αποκάλυψε ότι το πρόβλημα είναι ενδεχομένως ευρύτερο. Οπότε πήραμε και άλλα στοιχεία από τους καταγγέλλοντες και τους αναφέροντες, εκτός από αυτούς που είναι παρόντες. Και στην παρούσα φάση των διαδικασιών εξετάζομαι την, ε, από ό,τι φαίνεται, έλλειψη ε, δυνατότητας ένδικων μέσων σε αυτή την περίπτωση σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού όχι μόνο το, του ATA, αλλά όλων των κατηγοριών στα σχολεία τα δημόσια. Και φαίνεται ότι υπάρχει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση στους... Ε, λιγότερη, λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση σε αυτούς που είναι το του ορισμένου χρόνου. Αυτές οι διαδικασίες επί παραβάση δεν θα ε, έχουν άμεση ε, επικούρηση γιατί δεν παρεμβαίνει η Κομισιόν σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Όσοι νιώθουν ότι ε, υπέστησαν βλάβη θα πρέπει να προσφύγουν στα δικαστήρια της χώρας τους. Τώρα για ένα δεύτερο θέμα υπενθυμίζω στους αναφέροντες ότι η οδηγία η σχετική δεν προβλέπει την μετατροπή καταχρηστικών πρακτικών ε, συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Και για να το πω έτσι κάπως ε, διακριτικά, Υπάρχει εδώ πρόβλημα, αν πιέσουμε το θέμα της μετατροπής σε αορίστου χρόνου, ε, μπορεί να υπάρξει βλάβη. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι δεν αναφέρεται η μετατροπή από την οδηγία. Προβλέπει μόνο τη λήψη μέτρων και εμείς περιμένουμε να μας περιγραφούν τα μέτρα αυτά ποια θα είναι. Τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ιταλικών αρχών για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους στείλαμε τον Οκτώβριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μιράντα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να δηλώσω αλληλέγγυη με εκείνα τα πρόσωπα που σηκώθηκαν και ήρθαν εδώ. Τόσοι και τόσες από τους αναφέροντες. Και βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση ακριβώς όπως ε, προανέφεραν ε, και, καταδικάζουμε αυτήν την ασυνέπεια που τους ανάγκασαν να φτάσουν εκεί. Επίσης θα πρέπει να, να, να σας παραπέμψω στη, στην απόσταση 22 του 2012 και έχουμε αυτό το 385 εκεί αυτό το σημείο το οποίο μιλάει για αυτό το πρόβλημα. Εκεί ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι με προσωρινή σύμβαση εργασία ε, ή με μερική απασχόληση ε, είναι σε δημιουργική θέση σε σχέση με αυτού που εργάζονται σε πλήρη απασχόληση. Και έχουμε αυτέ τι δύο περιπτώσει Οπότε έχουμε αυτή, αυτή την ε, περίπτωση που έχουμε τη δυσμενή διάκριση βάρο αυτή τη εργαζομένη από την Ισπανία, η οποία ακριβώ παραπέμπει σε ε, αυτό, αυτό το χαρακτήρα, αυτέ τι συνέπειε των, των, των ε, τέτοιων συμβάσεων εργασία και ακριβώ τι γίνεται. ε, ε πρόκειται για συμβάσει ορισμένου χρόνου το αντίθετο, δηλαδή το τι γίνεται με τι συμβάσει αορίου του χρόνου ή τέλο με κάποια μακροχρόνια συμβόλαια. Οπότε κάποιο έτσι έχει κάποιε δόσει στη ζωή του. Είναι αναλυθέ το ότι σε τέτοιε περιπτώσει ε, είναι το, το πρόβλημα είναι εδώ πέρα οι, ότι οι βουλευτές δεν παρίστανται πολύ. Αλλά τελικά φταίει η κοινωνική Ευρώπη. Θα πρέπει να τηρείται το κοινωνικό κεκτημένο και επίσης από πλευρά μα Όσον αφορά δηλαδή, τους πράσινους, θεωρούμε ότι θα πρέπει να μην ανοιχτεί αυτή η αναφορά, οπότε και θα διαβιβάσουμε στη συνέχεια ε, σε, σε άλλη συνεδρία για να εξεταστεί αυτή η αναφορά. Πρόεδρος, για παρακαλώ συντόμως γιατί θα πρέπει να τελειώσουμε. Σύντομα θα τα πω. Σωστά τα είπε η προηγούμενη ομιλήτρια. Πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει οδηγία σε σχέση με το πώς μετατρέπονται οι ορι... Ε, ορισμένους σε Κάποια στιγμή πρέπει να ολοκληρωθεί η σύμβαση ορισμένου χρόνου. Βλέπω εδώ 11 φορές, 7 φορές ανανεώθηκαν, 10 φορές ανανεώθηκαν, παρατάθηκαν. Είναι άδικο αυτό. Οπότε η γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγία που προλαμβάνει αυτά και τα εμποδίζει. Ενθαρρύνω τους αναφέρουσες να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό. Μπράβο στην Κομισιόν που κινήθηκε γρήγορα με τη διαδικασία επί παραβάση κατά της Ιταλίας και πρέπει βέβαια η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή, να ξανασυζητήσουμε, να δούμε τι έγινε. Τελική παρατήρηση. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ντροπή και είναι και τραγικό το Ιταλικό κράτος να παραβιάζει τις ευρωπαϊκές ε, νομοθεσίες. Δεν είναι εταιρεία, δεν είναι καμιά πολυεθνική αυτή, είναι ένα κράτος το οποίο ε, παραβιάζει ε, νομοθετήματα τα οποία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα ενέκρινε μαζί με τους άλλους. Μάλιστα. Έχουμε πρόβλημα χρόνου, πρέπει να ολοκληρώσουμε διαφορετικά θα φύγουν οι διερμηνείς. Όμως νομίζω ότι δεν υπάρχουν αμφιβολίες. Χρειάζεστε ένα λεπτό για να απαντήσετε μάλιστα. Ήθελα απλώς ε, να ρωτήσω οι προσφυγίτες στο εργατικό δικαστήριο για τη σταθεροποίηση της σχέσης ε, εργασίας για την κυρία Πισάρτα είτε η προσφυγή στο δικαστήριο του Λάτσιο για την οριζόντια κινητικότητα. Μήπως ε, θα μπορούσε η Επιτροπή να μας ενημερώσει εξαντλητικά για το τι ακριβώς κάνει το τελικό κράτος αυτά τα χρόνια. Εγώ υπογραμμίζω ότι το άρθρο 5.4 του νομοθετικού διατάγματος 368 του 2001 καθορίζει ότι ένα, μια, μια σύμβαση διάρκειας άνω των τριών ετών θεωρούνται ως αορίστου χρόνου εργασία. και αυτό προκύπτει από τη μεταφορά του κοινοτικού δικαίου στο ιστορικό δικαίου. Έτσι λοιπόν είναι παράλογο το ίδιο το κράτο το Ιταλικό να παραβιάσει ε, ουσιαστικά ένα κανόνα που το ίδιο μετέφερε στο ιστορικό δίκαιο για να σεβαστεί την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Μάλιστα, σα ευχαριστούμε. Πέρα από τι μεμονωμένε υποθέσει. ε, ε, ε αυτά μπορούν ουσιαστικά να γίνουν προσφυγέ ενώπιον των εθνικών αρμοδιών Εμεί, θα ασχοληθούμε με αυτή την αναφορά κρατώντας την ανοιχτή και κατόπιν ε, θα ακολουθηθεί η διαδικασία. Σήμερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν εξάντλησε με μία, μας παρουσίασε μία ενημέρωση καινοτόμο για όλους εμάς ότι έναντι της Ιταλίας ξεκίνησε μια διαδικασία επί παραβάση επειδή παραβιάστηκε αυτή η νομοθεσία στην οποία εσεί αναφερθήκατε. Αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν θα επιλύσει τη μία και μόνη υπόθεση αλλά θα πρέπει να θέσει την ε, Ιταλία, ε, θα πρέπει να κάνει την Ιταλία να σεβαστεί πραγματικά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μας δώσατε και την ευκαιρία να είμαστε οι πρώτοι που μάθαμε αυτή την είδηση. Δυστυχώς δεν μας τιμά. Δηλαδή η διαδικασία επί παραβάση κατά της Ιταλίας ε, για αυτές ε, τις συμβάσεις ε, ορισμένου χρόνου. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Να σας αναφέρω και κάτι σε σχέση με τις αναφορές που έχουμε στο τμήμα Β της ημερησίας διάταξης. Ζητήθηκε να μεταφορθεί το σημείο 18, το σημείο 38 και το σημείο 45 να συζητηθούν εκ νέου. Σας χαιρετίζω. Καληνύχτα σας.